Bonjour euh, Ας αρχίσουμε, σας παρακαλώ, με την έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Θα γίνουν δύο τροποποίησεις στην ημερήσια διάταξη. Υπάρχει ένα μικρό λάθος στην ε, ημερήσια διάταξη. Σε σχέση με το σημείο 14 δεν θα ψηφίσουμε την έκθεση για το χρηματοδοτικό μέσο, αλλά μόνο τις τροπολογίες. και νομίζω ότι είναι περίπου 600 χρονοβόρα διαδικασία και επίσης την εντολή διαπραγμάτευσης. Αυτή είναι η πρώτη τροποποίηση. Η δεύτερη αφορά την έκθεση της κυρίας Γκρές. Θα μας ε, παρουσιάσει την έκθεση της σήμερα και όχι αύριο. Υπάρχουν σχόλια. Όχι, άρα εγκρίνεται η μυρίσια διάταξη. Εγώ δεν έχω ανακοινώσει ως πρόεδρος. Η Κομισιόν μας ανέφερε ότι θα ήθελε να κάνει ανακοίνωση. Και δίνω το λόγο στην κυρία Ελέν Μπουργκάτ. Έχουμε δύο ανακοινώσεις. Μία πληροφόρηση για την κοινωνική προστασία, ανταλλαγή πληροφοριών. Θα σας, μάλλον σας εξήγησα τις Γενικές Κατευθυντήριες Γραμμές τον Ιούνιο και στις 20 Αυγούστου 2012 εγκρίθηκε με βάση τις Γενικές Κατευθυντήριες Γραμμές που σας είχα προαναφέρει. Πρόκειται για γενικές κατευθυντήριες γραμμές που διέπουν αυτό τον τομέα και ως προς τις ευρωπαϊκές ημερίδες ε, ανάπτυξης 16 και 17 Οκτωβρίου θα μας παρουσιάσει το θέμα η κυρία Κριστιαν Σιμών. Ο κύριος, με συγχωρείτε. Όπως σας είπα, οι ημερίδες θα λάβουν χώρα στις 16 και 17 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες. Φέτος αναμένουμε 5.000 συμμετέχοντες θα σταθούμε σε δύο γεγονότα. Τη World Food Day 16 και την καταπολέμηση και εξάλληψη της φτώχειας της 17. Το βασικό θέμα της ημερίδας ε, ανάπτυξης αφορά τη βιώσιμη ανάπτυξη θα μιλήσουμε για την ασφάλεια τροφίμων, τον δημόσιο τομέα και την ολοκληρωμένη ανάπτυξη, inclusive growth. Αυτά θα αφορούν τις ημερίδες, αυτά τα θέματα. Στον κατάλογο συμμετεχόντων προσκεκλημένων, εδώ έχετε ένα ξεχωριστό έγγραφο, θα έχουμε 10 επικεφαλής κρατών, 5 επιτρόπους, και του Υπουργούς Ανάπτυξης 9 κρατών μελών. Εάν επιθυμείτε περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να τις δείτε στην ιστοσελίδα μας για το πώς θα διενεργηθεί, πώς προβλέπονται οι μερίδες. Επίσης, το λεπτομερές πρόγραμμα υπάρχει στο διαδίκτυο. Θα έχουμε 22 πάνελ υψηλού επίπεδου και 28 project labs. Ξέρετε ότι οι έξι τελευταίες εκδόσεις αφορούν ε, ένα το λεγόμενο Village of Development όπου παρουσιάζουμε τις διάφορες δραστηριότητές μας. Φέτος αποφασίσαμε να μην υπάρξει αυτό το χωριό της ανάπτυξης, αλλά να γίνουν διάφορες εκδηλώσεις σε συγκεκριμένες αίθουσες, όπου οι φορείς ανάπτυξης θα υποβάλουν τις διάφορες δραστηριότητες τους ή θα κάνουν ενημερώσεις. Έτσι θα υπάρχει μεγαλύτερη διάδραση μεταξύ συμμετεχόντων και stakeholders. Επίσης, πέρα από τον υψηλό αριθμό συμμετεχόντων, θα ε, μεταδίδονται από το διαδίκτυο όλα τα πάνελ υψηλού επίπεδου. Άρα, όποιος έχει σύνδεση θα μπορεί να παρακολουθήσει αυτά τα πάνελ υψηλού επίπεδου. Επίσης, προβλέπονται διάφορες δραστηριότητες και εκδηλώσεις μία σειρά ε, διαλέξεων για την ανάπτυξη στο ULB και διάφορες εκδηλώσεις στον χώρο Σανγκόρ. Εν γέννη διάφορες εκδηλώσεις προβλέπονται σε συγκεκριμένους χώρους. Σας προσκαλώ όλους. Μπορείτε να εγγραφείτε μέσω διαδικτύου είναι πολύ σημαντικό και θα πρέπει να γίνει προεγγραφή διότι μόνο όσοι κάνουν εγγραφή μέσω διαδικτύου θα διαθέτουν ένα badge συμμετοχής. Επίσης ε, και πολλοί ευρωβουλευτές θα συμμετάσχουν όπως εσείς ε, κυρία μου φαντάζομαι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ εκ των προτέρων για την παρουσία σας. Ευχαριστώ. Τώρα δίνω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να απαντήσει στο ερώτημα του Keith Taylor, του συναδέλφου μας. Ο κύριος Μικαέλ Ντοσέτρη θα απαντήσει. Η ερώτηση έχει τρία τμήματα. Πρώτον, τι έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να διαπιστώσει κατά πόσον αυτές οι πράξεις ε, των δυνάμεων ε, αμήνης του Ισραήλ είναι νόμιμες. Αν έχει ζητηθεί αποζημίωση και πώς και τρίτον τι μέτρα έχει λάβει η ε, Επιτροπή για να βοηθήσει ε, τους δικαιούχους να ζητήσουν αποζημίωση. Η Κομισιόν έχει επανειλημμένως πει πως ε, θεωρεί πως ε, αυτές οι ζημιές και οι καταστροφές υποδομών που έχει βοηθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη της να κατασκευαστούν στι κατεχόμενε παλαισθηνιακέ περιοχές είναι απαράδεκτες το επαναφέρει στην ατζέντα του πολιτικού διάλογου με το Ισραήλ συχνά και σε όλα τα φόρα που προβλέπονται από τη Συμφωνία με το Ισραήλ. Στις 14 ε, Μαΐου 2012 στο ε, Φόρουμ με το Ισραήλ καλέσαμε το Ισραήλ να τηρήσει τις ε, υποχρεώσεις που προκύπτουν από το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο σε ό,τι αφορά τον Παλαιστινιακό πληθυσμό είτε στην Δυτική Όχθη ε, Γάζα, στη λόρια της Γάζας, όπου έχουν γίνει και περισσότερες καταστροφές. Ε, ζητούμε να απλοποιηθούν διαδικασίες για τη χορήγηση άδειας οικοδόμησης στους Παλαιστινίους ε, και η, να διευκολυνθεί η πρόσβασή του στο νερό, στο είδωρ κλπ. Επίσης ζητήσαμε το Ισραήλ να προστατεύει τις ευρωπαϊκές επενδύσεις στο μέλλον. Σε ό,τι αφορά τα μέτρα που έχουν ληφθεί προκειμένου να ζητήσουμε αποζημίωση. Ε, καταστήσαμε σαφές στο Ισραήλ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένει ε, οι υποδομές αυτές να προστατεύουν από πλευρά του Ισραήλ. Ε, χρησιμοποιούμε τη, το διπλωματική οδό για να διασφαλίσουμε την προστασία αυτών των υποδομών. Το πρόβλημα που έχουμε αντιμετωπίσει είναι ότι αυτές οι επενδύσεις έχουν ήδη ε, ε, μεταφερθεί ως ιδιοκτησία στους Παλαιστινίους, στους δικαιούχους και εμείς πλέον δεν είμαστε κάτοχοι αυτών των υποδομών. Ε, οπότε δεν μπορούμε να ζητήσουμε αποζημίωση νομικά. Παρ' όλα αυτά έχουμε εκδώσει νότα διαμαρτυρίας επανειλημμένως στο Υπουργείο Μήνες του Ισραήλ για καταστροφές τέτοιου τύπου και για project τα οποία και ιδιαίτερα για project για τα οποία δεν έχουν δοθεί ακόμα στους ε, δικαιούχους. Ε, το, ε, μία μόνο φορά έχουμε λάβει αποζημίωση ε, για εγκαταστάσεις οι οποίες είχαν καταστραφεί στην Γάζα σε επίθεση του Ισραηλινού στρατού. Άλλες φορές δεν έχουμε καν λάβει απάντηση. Πώς βοηθάμε τους δικαιούχους, ε, αυτό προσπαθούμε να κάνουμε είναι να εξάγουμε διδάγματα από το παρελθόν. Από τις δικές μας απογοητεύσεις. Οπότε η προγραμματική, περίοδος, η προγραμματική διαδικασία του 2012 περιλαμβάνει μέτρα για την περιοχή C των κατεχομένων, μεταξύ αυτών υποστήριξη των Παλαιστινικών Αρχών για ε, προγραμματισμό υποδομών και για κάποιε μικρές υποδομές. Επί τόπου η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αποφασίσει και είναι δεσμευμένη ε, να ε, δείξει η ποιότητα με το Ισραήλ χωρίς να είμαστε επιθετικοί. Οι Ισραηλοί έχουν δείξει ότι θέλουν να συνεργαστούν μαζί μας επί τόπου, οπότε προσπαθούμε να το εκμεταλλευτούμε. τα project στο μέλλον θα τα συντονίσουμε στο μέτρο δυνατό με τις Ισραηλινές αρχές ε, και θα διατηρήσουμε εμείς ε, την ιδιοκτησία ε, των υποδομών όσο, το δούμε, όσο μπορούμε περισσότερο. Ενδεχομένως θα μπορούσαμε μάλιστα ακόμα και μετά τη μεταφορά της, του ιδιοκτησιακού καθεστώτος, μεταβίωση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος, να έχουμε μια συνεργασία για να τους βοηθάμε. Ευχαριστώ. Well, thanks very much. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που μας λέτε. Και θα ήμουν ευγνώμων αν είχαμε μια γραπτή απάντηση από εσάς και ίσως μια σύνοψη όλων όσων μας είπατε. Γιατί πιστεύω ότι πρέπει να το εξετάσουμε προσεκτικά. Αναφέρατε την, ε, τον τομέα C, το, της θάλασσας, τον τομέα C, που είναι όντως πάρα πολύ σημαντικός ιδιαίτερα όσον αφορά την ε, κατασκευή του παράνομου τείχους από την πλευρά του Ισραήλ αν ξεκαθαρίσατε ότι αναμένατε προστασία για εγκαταστάσεις οι οποίες χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά δεν έγινε και πολύ πρόοδος. 30 εκατομμύρια κόστησε η ζημία αυτή που προκλήθηκε σε αυτά τα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση έργα. Όπως βλέπετε δεν λειτουργεί αυτό το σχέδιο και ρωτήσαμε συγκεκριμένα ποια νομικά μέτρα σκοπεύετε να λάβετε για αποζημίωση. Σίγουρα δεν αμφισβητεί κανείς την αιτία ε, της ε, ζημίας αυτή, αλλά πραγματικά δεν καταλαβαίνω γιατί δεν καταφέραμε μέχρι τώρα να επιδιώξουμε αποζημίωση στην περίπτωση αυτή. Μας είπατε ότι θέλετε να υιοθετήσετε μία ήπια προσέγγιση του Ισραήλ και σίγουρα είμαι υπέρ μιας τέτοιας προσέγγισης, όμως εάν έχει αποτέλεσμα. Όμως αυτή η προσέγγισή σας που είναι θετική και χωρίς αντιπαράθεση δεν έχει αποτελέσματα. Έχουμε 30 εκατομμύρια ευρώ ζημία, δεν έχουμε καμία νομική διεκδίκηση και ποια είναι η απάντηση, ποια είναι η λύση σας. Πώς θα απαντήσετε σε αυτό ή είστε μια χαρά με το να βλέπετε αυτά τα χρήματα να σπαταλώνται αδίκως. Αυτές τις λεπτομέρειες θέλω από εσάς και θέλω κάποια διαβεβαίωση ότι η κατάσταση αυτή χειρίζεται από ικανά χέρια. Σας ευχαριστώ πολύ. Ξαναδίνω το λόγο στην Επιτροπή σε σχέση με μία ενδεχόμενη γραπτή απάντηση όπως ζήτησε ο κύριος Τέιλορ. Βεβαίως, κανένα πρόβλημα. Μπορούμε να χορηγήσουμε γραπτή απάντηση σε σχέση με τα άλλα σημεία νομίζω ότι η Κομισιόν και τα κράτη-μέλη συμμερίζονται την ανησυχία των κρατών μελών. Δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις σε σχέση με αυτή την ε, σχέση, με αυτή τη διελκυστίνδα η οποία ισχύει και ίσως η απόδοση υποδομών σημαίνει ότι δεν υπάρχει ίσως ε, νομοθετικό πλαίσιο παρέμβασης. Γι' αυτό νομίζω ότι για τα μελλοντικά σχέδια θα πρέπει να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια έτσι ώστε να υπάρχει ένα, μια νομική βάση, ένα σαφές ε, καθεστώς. Δεν ξέρω κατά πόσο η ΕΕ θέλει κάτι να πει ως προς το άλλο σκέλος της ερώτησης, προσπαθούμε με τους Ισραηλινούς να υποβάλουμε μία ε, ολοκληρωμένη ενωσιακού τύπου απάντηση από τα κράτη-μέλη, έτσι ώστε να έχουμε ισχυρότερη φωνή. θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια καταρχήν να ε, ακολουθήσουμε τη διαδικασία του Ισραήλ χωρίς να προβάλλουμε δικαίωμα αρνησή κυρίας. Όταν μιλάμε για μικρές υποδομές ε, εννοούμε ότι θα ακολουθήσουμε τη διαδικασία προγραμματισμού. Εάν μετά από παρέλευση εύλογου χρονικού διαστήματος δεν δοθεί συνέχεια, Δηλαδή, μετά τους έξι μήνες θα θεωρήσουμε ότι υπάρχει σιωπηρή συνένεση να προχωρήσουμε με τις υποδομές. Ο κύριος Τέιλορ για ένα λεπτό. Μάλιστα. Θα το ξαναπώ. Θα ήμουν ευγνώμων να ακούσω ποια δράση προτείνετε. Μας λέτε ότι δεν γίνεται κάτι γρήγορα, αλλά αυτό που γίνεται γρήγορα είναι ότι από το 2001 και μετά γρήγορα είναι η καταστροφή project αξίας 30 εκατομμυρίων ευρώ που χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και είμαι σίγουρη ότι τα μέλη είναι είναι εκνευρισμένα γι' αυτό και αναμένουμε από την Κομισιόν να αναλάβει κάποια δράση, να κάνει κάτι. Δεν μας έχετε πει αυτό που σκοπεύετε να κάνετε. δεν μας έχετε αναφέρει καμία θετική δράση και ελπίζω να προκύψει κάτι θετικό. Ευχαριστώ. Τώρα περνάμε στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης που είναι η έκθεση της Αντιπροέδρου μας, της κυρίας Ζανίκη για το πρόγραμμα Έρασμος για όλους. Πρόκειται για μία πρόταση ενός προγράμματος εκπαιδευτικού ε, χαρακτήρα κατάρτισης νεότητας και αθλητισμού που να απευθύνεται σε όλους και θα ήθελα να δώσω το λόγο στην κυρία Τζανίκη για να μας ε, υποβάλει τις τροπολογίες που προτείνονται στην έκθεση, την έκθεση Επιτροπής Πολιτισμού. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Το Νοέμβριο 2011 η Επιτροπή υπέβαλε ένα σχέδιο κανονισμού για τον έρασμο για όλους. Επρόκειτο για ένα πολιετές πρόγραμμα για τους νέους και τον αθλητισμό. Θέλουμε λοιπόν να ενώσουμε τις δράσεις στον τομέα αυτό μέσα στα πλαίσια ενός ενίου προγράμματος 2014-2020. Η Επιτροπή Πολιτισμού είναι υπεύθυνη, αλλά ζήτησε από την Επιτροπή μας να γνωμοδοτήσουμε επί της ουσίας. Ως ε, εισηγήτρια θα σας μιλήσω για τις σχετικές τροπολογίες για να γνωρίζετε καλύτερα το πλαίσιο. Το πρόγραμμα Έρασμος για όλους αναφέρεται στις πρωτοβουλίες και δραστηριότητες που αφορούν τον τομέα εκπαίδευσης. Και σε αυτά τα πλαίσια λαμβάνουμε υπόψη τον διεθνή χαρακτήρα συνεργασίας μέσα στα πλαίσια της τριτοβάθμιας εκπαίδευση, που είναι ύψη τη σημασία για την ε, έκθεσή μας, για την Επιτροπή μας, με συγχωρείτε. Θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει να προωθήσουμε αυτές τις δράσεις και να τις συγχωνεύσουμε σε ένα ενίο πρόγραμμα για να είναι πιο αποδοτικές και διαφανείς. Γι' αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να δεχτούμε τη σύσταση αυτή. Πέρα από αυτές τις ε, πρωταρχικές ε, υποδείξεις, μετά από εξέταση της έκθεσης ΠΑΚ, θεωρώ ότι στην πρόταση κανονισμού υπάρχει περιορισμένη μνήμα στις δράσεις που πρέπει να χρηματοδοτηθούν μέσω του DCI, του μας. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να ενισχύσουμε μηχανισμούς όπου εμπίπτουν αυτές οι δράσεις μέσα στα πλαίσια της αναπτυξιακής βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, ε, θεωρούμε ότι η χρηματοδότηση του DCI, του ΜΑΣ, δεν ε, αντιστοιχεί στο κριτήριο της δημόσιας ε, βοήθειας για αναπτυξιακούς σκοπούς, όπως ορίζεται στο 2014-2020. Ως προς τις τροπολογίες επί του σχεδίου ΠΑΚ έχω υποβάλει μία πρόταση και ζητώ την υποστήριξή σας. Χωρίς να μπω τώρα σε λεπτομέρειες, θα ήθελα να σας μιλήσω για τους στόχους των ε, τροπολογιών. Θέλουμε μία καλύτερη διάρθρωση των αναπτυξιακών στόχων για την καταπολέμηση της φτώχειας. Επίσης, να μιλήσουμε για μηχανισμούς κινητικότητας για να μην υπάρχει ε, για να μην υπάρχουν διαρροές εγκεφάλων. Επίσης, να υλοποιηθούν οι δράσεις σε πλήρη συμφωνία με τα αντίστοιχα μέσα, από τα οποία αντλούνται τα κονδύλια. Επίσης, θα πρέπει να οικειοποιηθούν τα προγράμματα τα κράτη-μέλη και να γίνει μια αποτίμηση έτσι ώστε να διασφαλίσουμε την ποιοτική αποτίμηση μέσα στα πλαίσια της διαφάνειας. Ίσως φαίνονται τεχνική υφής αυτές οι προδιαγραφές, όμως έχουν μεγάλη σημασία για την Επιτροπή μας. Στόχος αυτών των τροπολογιών είναι να υποστηρίξουμε τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανάπτυξη και χρηματοδότηση μέσα στα πλαίσια του νέου μας και να δράσουμε τάχιστα υπέρ των χωρών που το χρειάζονται. Θα πρέπει λοιπόν να υποστηρίξουμε αυτές τις αρχές σε όλους τους τομείς και περιμένω τα σχόλιά σας επί των τροπολογιών όπως έχουν διαμορφωθεί. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Γκρέσ έχει το λόγο. Καλή σας μέρα. Θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Ζανούκη. Εξ ονόματος της ομάδας των Πρασίνων, εν γέννη, συμφωνούμε με την προσέγγιση της. Καταρχήν ε, το πρόγραμμα Εράσμος για όλους προβλέπει ε, ε, χρηματοδότηση για τους νέους και με μάλιστα με νέο τρόπο και αυτό είναι πολύ καλό. Ο κίνδυνος είναι βέβαια να χαθεί η ταυτότητα του καθόλου από τα προγράμματα τα οποία εντάσσονται πλέον στο Εράσμος για όλους. Ε, και να επικρατεί σύγχυση μεταξύ των δικαιούχων. Ε, και σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση της φτώχειας, ε, θέλουμε να υποστηρίξουμε την εισηγήτρια. Η σύνδεση ανάμεσα στο σχέδιο κανονισμού και στα μέσα χρηματοδότηση για την ανάπτυξη, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξη για παράδειγμα, πρέπει να γίνει σαφής. Επίσης, συμφωνούμε με την ε, ανάγκη να γίνουν σεβαστές οι διαδικασίες των διαφόρων μέσων και βέβαια οι αρμοδιότητες ελέγχου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τρίτον, συμφωνούμε επίσης με την ανάγκη η χρηματοδότηση να γίνει επί τη βάση μιας πολυε... ενός πολιετούς προγραμματισμού με βάση άξονες προτεραιότητας που θα καθορίζονται από τις συγκεκριμένες ενδιαφερόμενες χώρες. Παρ' όλα αυτά, θα μπορούσαμε ενδεχομένω να πάμε λίγο πιο μακριά. Πώς? Ε, είναι απολύτω αναγκαίο να γίνεται έλεγχο εκ των προτέρων για να αποφύγουμε αυτό που είχαμε πάθει πριν από λίγο καιρό με τον κύριο Γκέρεντς με τη Βραζιλία, θυμάστε, με το ε, μηχανισμό αναπτυξιακής συνεργασίας ε, γιατί τότε θυμάστε ότι ε, η ε, επιδοτήσεις ε, υποτροφίες του έρασμους ε, πηγαίναν σε πλούσιες οικογένειες που έστελναν τα παιδιά τους να σπουδάσουν στην Ευρώπη. Λοιπόν, θέλουμε να το αποφύγουμε αυτό. Θέλουμε να φτάνουν τα κονδύλια σε ανθρώπους που πραγματικά τα έχουν ανάγκη. Τέλος, θα ήθελα να συμφωνήσω με το θέμα της πρέπει να αποφύγουμε τη διαρροή εγκεφάλων, όπως είπατε. Ευχαριστώ. Κύριος Γκέραντς. <clears throat> Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω με τη σειρά μου την κυρία Τζανίκη για την εισήγησή της. Είναι αρκετά επικριτική η έκθεσή της και θα ήθελα να σταθώ στο θέμα της χρηματοδότησης γιατί μιλάτε για την ε, δυνατότητα ολοκλήρωσης της διαδικασίας. Από την άλλη όμως, θεωρείται ότι οι συντάκτες του κειμένου δεν είναι και τόσο συνεπείς. Αντιφάσκουν. Και θα ήθελα να ρωτήσω ιδιαίτερα την ε, Κομισιόν τι θα αναλάβει ο μηχανισμός και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης ε, θα συμμετάσχει στο Erasmus Mundus. Η συγγήτρια πολύ σωστά μιλάει για τη συμβατότητα του χρηματοδοτικού σκέλους της ΕΤΕ ή του ΜΑΣ μέσα στα πλαίσια της ένταξης στην διαδικασία αυτή. Μπορείτε να μας εξασφαλίσετε ότι τα χρήματα αυτά που θα χορηγηθούν για το μηχανισμό αναπτυξιακής συνεργασίας θα έχουν όλες τις ρήτρες διασφάλισης Επίσης, ζητήσαμε να υπάρξει αντιστάθμιση του μας μέσα στα πλαίσια της ε, ανάκαμψης της κατάστασης, διότι τι κάνουμε, αντλούμε από διάφορα τμήματα, αλλά είχαμε τις δικές μας απόψεις πριν από την Κομισιόν σε σχέση με τον όγκο συναλλαγών του ΜΑΣ. Δηλαδή, λάβαμε υπόψη και το μυς της στήλη 4 ως προς την αιρεσιμότητα. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Θα χρηματοδοτήσουμε την κατάρτιση στις υποανάπτυξη χώρες από το Μηχανισμό Αναπτυξιακής Συνεργασίας αυτό θα πρέπει, αυτό θα πρέπει να είναι επικερδές, όπως είπε και η κυρία Γκρές, για τις υποανάπτυξη χώρες. Θα πρέπει να υπάρχει όμως η αρχή της αιρεσιμότητας, δηλαδή ρήτρε διασφάλισης. Ας πούμε καταρτίζουμε ε, ιατρούς εχεί χρόνια. Τι εγγύησεις έχουμε ότι τα προγράμματα, τα χρήματα αυτά θα, χρησιμοποιηθούν για χι χρόνια για τους συγκεκριμένους ιατρούς, για τη συγκεκριμένη κατάρτιση, που ξέρουμε ότι δεν θα χρησιμοποιηθούν αλλού. Πώς μπορεί να υπάρχει αιτιώδη συνάφεια, δηλαδή μεταξύ της χορήγησης αυτών των χρημάτων και των υποτροφιών των συγκεκριμένων, όπου ε, οι γιατροί στη συνέχεια με βάση τους οποίους μηχανισμούς οι γιατροί στη συνέχεια θα υπηρετήσουν στις χώρες τους, στη χώρα προέλευσης. Θα πρέπει έτσι να αποφύγουμε τη διαρροή εγκεφάλων που πολλές φορές θίγουμε χωρίς να βλέπουμε πάντα τις συνέπειες. Το λόγο έχει επιτροπή. Η κυρία Κλέρ Μαντέλ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ όλα τα μέλη τα οποία βοήθησαν σε αυτή την θετική μάλλον γνωμοδότηση. Στόχος της Κομισιόν όπως γνωρίζετε είναι να βάλει κάτω από την ίδια ομπρέλα όλα τα υπάρχοντα προγράμματα τα οποία ε, είναι κατακαιρματισμένα αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν ε, πολλά που καλύπτουν το ένα τη Λατινική Αμερική, το άλλο τι γειτονικέ μας χώρες, ένα άλλο την Αφρική, ένα άλλο την τριτοβάθμια εκπαίδευση, ε, το Erasmus που καλύπτει ε, την κινητικότητα των ε, φοιτητών και του ακαδημαϊκού προσωπικού. Οπότε η πρόταση ήταν και είναι όλα αυτά να καλυφθούν από το ίδιο πρόγραμμα, να μπουν στην ίδια ομπρέλα και να ενοποιηθούν έτσι ώστε να ενισχυθεί και η σύνδεση ανάμεσα στο ευρωπαϊκό και το διεθνές. Δηλαδή υπάρχει το πρόγραμμα της διαβίου μάθησης, που, του οποίου το κομμάτι της ανώτερης της εκπαίδευσης είναι το έρασμος και από την άλλη μεριά υπάρχει το έρασμος μούντους. Ε, θέλουμε αυτά τα δύο για παράδειγμα να τα βάλουμε μαζί και να τα συνδέσουμε. Ε, έχουμε στον τομέα 1 και στον τομέα 4 δύο διαφορετικές χρηματοδοτήσεις. Πρότασή μας είναι αυτή τη στιγμή δηλαδή να... Ε, έχουμε διπλή χρηματοδότηση, το 80-90% του προγράμματος ε, από τον τομέα 1 και το υπόλοιπο 10-20% από τον τομέα 4, τα 5 δηλαδή μέσα τα οποία αναφέρατε. Ε, ε, το, το ΜΑΣ, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης και, το, και την πολιτική γειτονίας η επταετής περίοδος από την άλλη μεριά προβλέπεται ε, είναι πολύ παρόμοια με αυτή που είχαμε ήδη προβλέψει ως τώρα στις δράσεις συνεργασίας μας ε, στα έτη 2013. Ε, Συνεπώς η αύξηση τελικά δεν είναι πολύ μεγάλη, είναι 10%. Ζητούμε λοιπόν χρηματοδότηση και από τον τομέα 4, οπότε είναι προφανές πως η χρηματοδότηση από το Μηχανισμό Αναψυχιακής Συνεργασίας ε, θα μπορέσει να αφιερωθεί μόνο σε δράσεις συνεργασίας για την κινητικότητα ε, με δικαιούχους συγκεκριμένης περιοχής. Καταλαβαίνουμε επίσης ότι θα πρέπει να σεβαστούμε τους στόχους του καθενός από αυτά τα μέσα. Άλλωστε αυτό συμβαίνει και τώρα ήδη. Το Erasmus Μούντους για παράδειγμα χρηματοδοτείται ήδη από πέντε μέσα και λειτουργεί πολύ καλά σεβόμαστε κάθε φορά τους στόχους του κάθε ε, μέσου που χρησιμοποιούμε το ίδιο θα συμβεί και με, με τον προγραμματισμό είναι δύσκολο να έχουμε πρόγραμμα που να καλύπτει όλο τον κόσμο ε, και ε, να είναι και να το διαπραγματευτούμε με κάθε μία από τις ε, χώρες ε, ξεχωριστά. Θα έχουμε όμως περιφερειακό προγραμματισμό, ένα φόρουμ αναπεριφέρεια όπου θα διαβουλευόμαστε με τους ενδιαφερόμενους. Τώρα να απαντήσω σε ορισμένα προβλήματα τα οποία αναφέρθηκαν. Προκειμένου τα ευρωπαϊκά και μη ευρωπαϊκά πανεπιστήμια να ε, έχουν να είναι προβλέψη, να έχουμε μια προβλέψιμη χρηματοδότηση. Ε, έχουμε ε, προβλέψει ε, όπως μας ζήτησαν κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης Ο προγραμματισμός να γίνεται για περίοδους 3-4 ετών. Αυτό μας ζήτησαν τα Ιδρύματα. Από την άλλη μεριά Ε, όπως σας είπα, ο πραγματισμός γίνεται σε περιφερειακό επίπεδο, σεβόμαστε ε, τους κανονισμούς των διαφορών μέσων, ε, θα πρέπει να υπάρχει οπωσδήποτε μια διάσταση ανάπτυξης, υπάρχει μια πτυχή κινητικότητα, αλλά δεν είναι η μόνη, υπάρχει κινητικότητα για του φοιτητέ, για το ακαδημαϊκό προσωπικό, αλλά ένα μεγάλο κομμάτι του προγράμματο θα είναι το capacity building, το ονομαζόμενο capacity building, ε, δηλαδή η βοήθεια προς τα πανεπιστήμια στο, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης να εξυγχρονιστούν, να αναπτύξουν ε, προγράμματα, ε, εκπαιδευτικά προγράμματά τους κλπ. Σε ό,τι αφορά τι θετικέ διακρίσει, είναι προφανέ ότι αν έχουμε δύο φοιτητέ του ίδιου επίπεδου, πάντοτε θα δίνουμε προτεραιότητα σε αυτόν τον φοιτητή που προέρχεται από τι πιο ε, άπορες, από την πιο άπορη οικογένεια. Το ίδιο κάνουμε και στο έρασμο, στο εσωτερικό, ε, σε ακαδημαϊκό επίπεδο, σε επίσδιο ακαδημαϊκό επίπεδο, επίδιο, σε επίδοση, σε πάντοτε δίνουν προτεραιότητα στους λιγότερο ε, ε, πλούσιους. Ε, μην ξεχνάτε ότι αυτή η συνεργασία υπάρχει πολύ συχνά εδώ και πολύ χρόνο. Ε, εδώ και 20 χρόνια λειτουργούν ορισμένα από αυτά τα μέσα ε, και πρόκειται να δώσουμε μια συνέχεια λοιπόν σε αυτούς τους μηχανισμούς που έχουν και τις δικές τους, ε, σε αυτές τις συνεργασίες που έχουν και τους δικούς τους μηχανισμούς διαβούλευσης. Σε ό,τι αφορά τον περιφερειακό προγραμματισμό και την περιφερειακή συνεργασία, μιλάμε για κονσόρσια πανεπιστημίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε διάφορες περιοχές του κόσμου και θα τους ζητήσουμε να μας υποδείξουν ή τα ίδια τις προτεραιότητές τους σε περιφερειακό επίπεδο. Έχουμε για παράδειγμα σε κάθε μία από τις χώρες γραφεία συντονισμού στα οποία λαμβάνει χώρα, ε, λαμβάνει χώρα διαβούλευση με τα αντίστοιχα υπουργεία της χώρας και πρόκειται να συνεχίσουμε να χρηματοδοτούμε αυτά τα δίκτυα. Νομίζω ότι κάλυψα όλα τα ζητήματα που εφηγήσαν. Παρ' όλα αυτά, αν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις, θα απαντήσω με τα χαρά. Ο κύριος Γκέρενς έχει το λόγο. Δεν ξέρω αν κατάλαβα καλά όλους τους όρους της αιρεσιμότητας. Δεν ξέρω αν απάντησε καν η Κομισιόν επί του θέματος. Oui. Alors η Επιτροπή. Όπως σας είπα, υπάρχει ένας διαθεσμικός χαρακτήρας στον έρασμο για όλους, δηλαδή δεν θα χρηματοδοτήσουμε την κινητικότητα όλων των φοιτητών. Για να μπορέσει ένας φοιτητής να ευεργετηθεί από την κινητικότητα θα πρέπει να υπάρχει εταιρική σχέση, συνεργασία μάλλον, μεταξύ δύο πανεπιστημίων να υπάρχει ένα learning agreement, μία συμφωνία μάθησης με συγκεκριμένες διευκρινήσεις για το τι αναμένεται από κάθε φοιτητή. Έτσι ώστε να είναι υπόλογος ο φοιτητής στο ίδρυμα από όπου προέρχεται. Και μόνο τότε μπορεί να τύχει χρηματοδότησης. Γκέρενς. Άρα Άλλο θα ήθελα να ξέρω, ορίζετε κανόνες για να, μην, για να αρνηθείτε τη συνεργασία, τη θεσμική συνεργασία μεταξύ ε, πανεπιστημίων. Δηλαδή, πώς μπορείτε να πείτε γιατί λέτε όχι σε δύο πανεπιστήμια μέσα στα πλαίσια της ε, δημόσιας, των δημόσιων χορηγήσεων και επιδοτήσεων. Τους κανόνες του DAX τους έχουμε ορίσει λεπτομερώς μέσα στα πλαίσια του capacity building. Πρόκειται για δραστηριότητες που προβλέπονται από το DAC. Τα πανεπιστήμια θα πρέπει να απαντήσουν σε εκδηλώσεις ενδιαφέροντος όπως ισχύει τώρα. Και αν τα πανεπιστήμια δεν τηρούν αυτούς τους όρους, δεν θα μπορέσουμε να τα δεχτούμε. Ως προς την κινητικότητα, την κινητικότητα των φοιτητών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν υπάρχουν ε, προβλήματα με το πρόγραμμα DAC. Το πρόβλημα αφορά περισσότερο τους φοιτητές και το προσωπικό που θέλουν, που μάλλον βρίσκονται εκτός μας ή στο τέλος του DCI. Αυτό το θέμα είχε ήδη φύγει μέσα στα πλαίσια του Erasmus Mundus. Μέσα στα πλαίσια της εκπαίδευσης και του πολιτισμού θέλουμε να αποστέλλονται φοιτητέ και διδακτικό προσωπικό στις υποανάπτυξη χώρες για να μην υπάρχει διαρροή εγκεφάλων. Άρα να γνωρίζουν καλά την κατάσταση όπως επικρατεί στον αναπτυσσόμενο κόσμο και θεωρούμε ότι αυτή η κινητικότητα προς τα έξω δεν μπορεί να υποστηριχτεί από τον μας θα πρέπει να βρούμε άλλους τρόπους χρηματοδότησης αυτής της προς τα έξω κινητικότητας. Εδώ μόνο υπάρχει πρόβλημα συμβατότητας, διαφορετικά για την κατάρτιση του διδακτικού προσωπικού, για τον εξοπλισμό των πανεπιστημίων, για την κινητικότητα του διδακτικού προσωπικού μέσα στα πλαίσια της κατάρτισης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δεν νομίζω ότι υπάρχει πρόβλημα συμβατότητας. Η κυρία Τζανίκη, ε, λυπάμαι γιατί καθυστερήσαμε και θα πρέπει να σας διακόπτω μετά από λίγα λεπτά. Ευχαριστώ. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω τη Γραμματεία της Επιτροπής μας για την υποστήριξη κατά την σύνταξη αυτής της γνωμοδότησης και τους συναδέλφους που παρενέβησαν σήμερα. Είναι πολύ σημαντικό το πρόγραμμα Έρασμος για όλους. Επίσης, είδα ότι σας απασχολεί το ζήτημα και θα ήθελα να σας πω ότι στις 20 Σεπτεμβρίου είναι η προθεσμία υποβολής τροπολογιών. Μην το ξεχνάτε αυτό, 20 Σεπτεμβρίου. Νομίζω λοιπόν ότι το πρόγραμμα Έρασμος για όλους αποτελεί ε, έναν φορέα μετάδοσης πολιτισμού και αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς την κατάρτιση. Σας ε, υπενθυμίζω ότι η προθεσμία υποβολής τροπολογιών είναι η 19 Σεπτεμβρίου στις 12 το μεσημέρι και Α, με συγχωρείτε, λέει πρόεδρο, έκανα λάθο. Όχι, 20 Σεπτεμβρίου, 20 Σεπτεμβρίου, όπως μας είπε και η εισηγήτρια, στις 5 το απόγευμα. Και η ψηφοφορία θα διεξαχθεί στις 9 Οκτωβρίου. Περνάμε στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης σε σχέση με μία αλλιευτική συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Γρυλανδίας που εξαρτάται από την κυβέρνηση της Δανίας. Η συντάκτριά μας είναι η κυρία Μάισνερ, στην οποία και δίνω το λόγο για να μας μιλήσει για το χρηματοοικονομικό πλαίσιο και τους άλλους όρους που διέπουν αυτή τη συμφωνία. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε έχουμε να κάνουμε με μια σύμπραξη ελληνική συνεργασία ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την κυβέρνηση της Δανίας και την, ε, κυβέρνηση της Χρυλανδίας. Επί της ουσίας υπευθύνη είναι η Επιτροπή Αλληλείας και ο συναδέλφος Όλε Κρίστενσεν. Η Γρυλανδία είναι μία από τις ήχε ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην περίπτωση αυτή είναι πάρα πολύ σημαντικό σημαντικό ε, για την Γρυλανδία, διότι ο τομέας της αλληλεία, ισοδυναμεί με 32% του ΑΕΠ της χώρας. Είναι δηλαδή το πιο σημαντικό έσοδο για την οικονομία της χώρας. 88% των ταπανών της Γρυλανδίας, των εξαγωγών της Γρυλανδίας ε, πηγαίνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι προϊόντα ε, αλληλείας. Για εμάς ως Επιτροπή Ανάπτυξης είναι σημαντικό αυτή η σύμπραξη ελευτική συνεργασίας να παραμείνει όσο έχει να υπαχθεί στα πλαίσια της ε, κοινής πολιτική πολιτικής και να συνδεθεί και με την σύμπραξη που έχουμε με την Γρυλανδία. Η σύμπραξη αυτή θα διαρκέσει μέχρι το 2013, άρχισε το 2007 και πρέπει να διασφαλιστεί ε, η ομαλή συνέχειά της. Ε, ε, η συμφωνία που έχουμε με την Γρυλανδία τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου του 2007 και 31 Δεκεμβρίου του 2012, φέτος δηλαδή, λίγη μετά από το εξαετές πρωτόκολλο και προβλέπεται επιμήκυνση για τρία άλλα χρόνια. Για, σε αυτό το πρωτόκολλο συμπεριλαμβάνονται και παράδειγμα οι ενισχύσεις, οι τα αλλιεύματα και το συνολικό ύψος των αλλιεύματων που θα αλλιεύονται και οι το μεγαλύτερο μέρος της επιχορήγησης πηγαίνει στα αλλιεύματα και ένα άλλο μέρος στις, στις υποδομές, ε, τις αλλιευτικές υποδομές. Τα αλλιεύματα βρίσκονται μονίμως υπό έλεγχο και φυσικά θέλουμε να υποστηρίξουμε την βιώσιμη αλία, ιδιαίτερα όσον αφορά τον, την υπόγλωσσα της Γρυλανδίας το, και τον Γάδο, τα οποία έχουν χαμηλούς πληθυσμούς, ε, εκεί πρέπει να θέσουμε πιο χαμηλά όρια. Σε γενικές γραμμές ε, υποστηρίζω την ε, συμφωνία του Κοινοβουλίου για την απέκταση της συμφωνίας αυτής τονίζοντας βέβαια ως κύριο σημείο των ε, ενδιαφερόντων μας την βιώσιμη αλία και τη διασφάλιση αυτής, ιδιαίτερα για τα ε, είδη που απειλούνται, την υπόγλωσσα της Γρυλανδίας δηλαδή, τον γάδο και τα κοκκινόψαρα. Επίσης πρέπει να φροντίσουμε για διαφάνεια και συνοχή με την αναπτυξιακή πολιτική. Τέλος, πρέπει να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα προκειμένου να αυξηθεί ο αριθμός των ελιμενισμών των ευρωπαϊκών σκαφών σε λιμένες της Γρυλανδίας με στόχο την τόνωση της ε, τοπικής απασχόλησης και των επιχειρηματικών ευκαιριών. Ε, να πω κλείνοντας ότι οι προθεσμίες πρέπει να κατατεθούν μέχρι την Τετάρτη, μέχρι τις 19. Ξέρω ότι είναι πολύ μικρό το χρονικό περιθώριο, όμως μόνο έτσι θα διασφαλιστεί ότι μέχρι το τέλος του χρόνου θα μπορούμε να υιοθετήσουμε τη νέα συμφωνία, έτσι ώστε να ισχύσει, να τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του 2013. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριος Αρσένης. Uh, Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ. Είναι μια σπάνια περίπτωση συμφωνίας αλλιευτικής σύμπραξης όπου παρατηρούνται τα παρατηρείται πολύ ομαλή εξέλιξη. Έχουμε δύο, τρία είδη που υπερελιεύονται, ο γάδος, η υπόγλωσσα της Γρυλανδίας και το κοκκινόψαρο. Αλλά πέραν αυτών η κατάσταση έχει ως εξή Τα επίπεδα των αλλιευμάτων ε, καθορίζονται βάσει επιστημονικών μελετών. Η μείωση των αλλιευτικών ευκαιριών για τα αλλιεύματα είναι σύμφωνα με τις συστάσεις και επίσης υπάρχει μια επιτροπή η οποία ελέγχει την εφαρμογή των, των ε, αληφτικών συμπράξεων και επίσης υπάρχει και μία ρήτρα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αυτό είναι κάτι το οποίο ζητούμε πάντα Βέβαια η Γρυλανδία δεν είναι αναπτυσσόμενη χώρα φυσικά. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε και άριστες εγγύησεις για τον σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Σε γενικές γραμμές πιστεύω πως δεν ήταν απόλυτα αναγκαίο για αυτήν εδώ την Επιτροπή να συντάξει γνωμοδότηση για το συγκεκριμένο θέμα, όμως εξακολουθεί να είναι κάτι πάρα πολύ επίγον, ιδιαίτερα για τις υπόλοιπες ανα... για τις υπόλοιπες αναλύσεις του δυνητικού πληθυσμού και που είναι άλλωστε και πολύ σημαντικό για το περιβάλλον. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι όντω η Επιτροπή Ελίας είναι η επί της ουσίας αρμόδια για αυτό το θέμα. Πιστεύω πως οι γενικές γραμμές είναι μια καλή ανάλυση δυνητικού πληθυσμού, η ανάλυση που έχει γίνει για τα αλλιεύματα αυτά και πραγματικά εύχομαι και οι επόμενες παρόμοιες αναλύσεις να είναι τόσο καλές όσο αυτή. Ευχαριστώ πολύ κυρία Λαβίν, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Μάισνερ, για την έκθεσή σας. Ε, μια έκθεση που βρίσκω πολύ καλή, ιδιαίτερα όσον αφορά την έκθεση αξιολόγησης. Συμφωνώ με τον κύριο Αρσένη Όντω, ε, γιατί η Επιτροπή ανάπτυξη να συντάξει γνωμοδότηση για την Συμφωνία Ελληνική σύμπραξη Ευρωπαϊκή Ένωση Γρυλανδία. Σίγουρα η Γρυλανδία, ναι, δεν είναι αναπτυσσόμενη χώρα. Βέβαια, η Κομισιόν θα μα το απαντήσει αυτό καλύτερα. Ωστόσο, δεν συμφωνώ πολύ με τον κύριο Αρσένη για το ότι αυτή είναι μια πρότυπη συμφωνία την οποία θα πρέπει σίγουρα να στηρίξουμε, διότι Πιστεύω πως η απόλυτη και θεμελιώδης αρχή που πρέπει να ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλες τις παρόμοιες συμφωνίες ελευτικής σύμπραξης είναι να μην συνεισφέρει στην εκμετάλλευση στην υπερ... Ε, των αλλιευμάτων, στην υπεραλίευση. Όντω όπως αναφέρθηκε, αυτά τα αλλιεύματα, τα τρία αυτά ψάρια υπεραλλιεύονται, ο γάδο, το κοκκινόψαρο και η υπόγλωσσα τη Γρυλανδία. Και με ανησυχεί πάρα πολύ ε, αυτό που διαβάζω από την ISIS. Αν αρχίσουμε με την υπόγλωσσα της Γρυλανδίας, θα δούμε ότι τα αποθέματα είναι, έχουν άγνωστο αριθμό. Δεν υπάρχει σχέδιο διαχείρισης. Ωστόσο, η ISIS συμβουλεύει ότι δεν θα πρέπει να λιεύονται πάνω από 8.000 τόνοι ετησίω, όμω τώρα αυτό που, το ποσό που ισχύει είναι 15.000 τόνοι ετησίω, πάνω από το σχεδόν το διπλάσιο δηλαδή. Θα μπορούσαμε λοιπόν να πούμε ότι υπάρχει ένα πλεόνασμα αυτών των αλλιευμάτων, στο οποίο έχει πρόσβαση η Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ η ανώτατα, τα επιτρεπτά όρια του, για το ψάρι αυτό είναι τα μισά. Όσον αφορά το ψάρο τώρα, το οποίο είναι ε, βενθικό είδος. Οι εκτιμήσεις που έχουμε αυτή τη στιγμή δείχνουν ότι οι αριθμοί του είναι οι χαμηλότεροι που έχουν παρατηρηθεί ποτέ και ο ρυθμός εκμετάλλευσης για το κοκκινόψερο είναι άγνωστος. Και τέλος για την υπόγλωσσα της Φιλανδίας. Υπάρχει ένα σχέδιο διαχείρισης ε, που αναπτύσσεται αυτή τη στιγμή. Και εδώ όμως είναι άγνωστος ο αριθμός της υπόγλωσσας της Γρυλανδίας και πάλι βλέπουμε ότι λείπουν πολλά, όπως και πριν δεν γνωρίζουν ακριβώς τον ρυθμό της εκμετάλλευσης της υπόγλωσσας της Γρυλανδίας. Αλλά πραγματικά φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή το, η υπόγλωσσα είναι στο 55% του BMSY από τα τέλη της δεκαετίας του 90. Αλήθεια, η Κομισιόν πιστεύει ότι αν υπάρχει μια πολιτική συμφωνία για ένα σχέδιο διαχείρισης ενός υπεραλλιευμένου είδους πραγματικά θα βοηθήσει, πραγματικά... Επίσης, αν δούμε τα ποσά, το σύνολο όλων αυτών των αλλιευμάτων, θα δούμε ότι πραγματικά ο ρυθμός είναι μεγάλος. Υπάρχει ο καπελάνος, για παράδειγμα, ένα βιομηχανικό είδος που αλλιεύεται με ρυθμούς 60.000 τόνων το χρόνο και φαίνεται ότι είναι ένα πολύ σημαντικό είδος για τον ε, ευρωπαϊκό στόλο. Διαφορετικά δεν θα γινόντουσαν διαπραγματεύσεις. Εγώ πιστεύω ότι δεν θα έπρεπε να μη συμπεριλαμβάνεται και αυτό το είδος, γιατί πάντα λέμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να προωθεί την βιώσιμη αλληλεία. Και αυτό είναι και... Και αυτό είναι και η ραχοκοκαλιά της, ε, των συμφωνιών αλληλευτικής σύμπραξης. είναι η συμφωνία αυτή πραγματικά συμβατή με την μη εκμετάλλευση ή πλεονάσματος εάν ο αριθμός του ελεύματος δεν είναι γνωστός ή εάν σύμφωνα με ε, επιστημονικές έρευνες το είδος αυτό υπεραλλιεύεται. Ευχαριστώ πολύ. Το λόγο έχει ο κύριος Πόγκα. Ευχαριστώ. Θα είμαι σύντομος. Θέλω να συγχαρώ την εισηγήτρια έλαβε υπόψη τα συμπεράσματα της ε, εκ των στέρων αξιολόγησης της ισχύουσας συμφωνίας και προτείνει την ε, ε, υιοθέτηση του καινούργιου πρωτοκόλου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενισχύει το τους δεσμούς της με τη Γρυλανδία με αυτόν τον τρόπο. Η Γρυλανδία είναι μία από τις 26 περιοχές και διαμερίσματα, υπερπόντια διαμερίσματα που συνδέονται με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Χαίρομαι γι' αυτό. Ευχαριστώ. Ο λόγος στην Κομισιόν. Thank you, Madam Chair. members, good afternoon. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σε όλους. Καταρχάς, να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την δουλειά και για την έκθεση σε αυτή τη Συμφωνία Αλληλευτικής Σύμπραξης και το, την ανανέωση του πρωτοκόλου. Όσον αφορά τη συμφωνία καθ' αυτή, δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, τις ξέρετε εξάλλου. Όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις με την Ιρλανδία, να πω ότι στο τέλος και οι δύο πλευρές εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για τα αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα τα οποία, όπως βλέπετε, σέβονται και τα δύο συμβαλόμενα μέρη και τονίζουν μία βιώσιμη προσέγγιση. Ιδιαίτερα, επίσης το πρωτόκολλο αυτό τονίζει την ε, στενή συνεργασία ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Γρυλανδία στην, στον τομέα της αλληλείας. Πολλά θέματα θίξατε, αγαπητά μέλη. Όντως, και πολύ σωστά αναφέρθηκε ότι υπάρχουν πολλές καινούργιες ρήτρε, ιδιαίτερα εκείνη που αναφέρεται στα ανθρώπινα δικαιώματα. Και αυτό είναι και το τυπικό που ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε, όλες τις παρόμοιες ε, συμφωνίες. Σε γενικές ε, γραμμές ακολουθήσαμε τις τα αποτελέσματα των ε, επιστημονικών μελετών όσον αφορά τα αλλιεύματα και σε σχέση με το παλιό πρωτόκολλο εδώ ε, βλέπουμε μία σημαντική μείωση στις ποσοστώσεις και για τα πελαγικά ψάρια και για, το, για την υπόγλωσσα της Ιρλανδίας. Για το κοκκινό ψαρό μειώθηκε, ήταν το διπλάσιο πριν. Για την υπόγλωσσα της Γρυλανδίας από περίπου 7.000 σε περίπου 3.000. 4.000 τόνους, με συγχωρείτε. Αυτές οι ποσοστώσεις είναι ενδεικτικές, δεν υπάρχουν στις, σε άλλες συμφωνίες. Η συγκεκριμένη συμφωνία προέκυψε μετά από ετήσιες ε, συναντήσεις. Και ακόμα και αν φαίνεται υψηλή αυτή η ποσόστοση, δεν είναι η τελική ποσόστοση για, τα, για το κάθε έτος που ακολουθεί. Ένα, τώρα ένας πιο λεπτομερής σχολιασμός για τα ληφτικά αποθέματα. Για αυτές τις τρεις νέες ποσοστώσεις ακολουθήσαμε μια πιο προσεκτική προσέγγιση και την ε, συμπεριλάβαμε και στο κείμενο. Για τον γάδο, όντως, εισήχθη πρόσφατα στο πρωτόκολλο η διασφάλιση της εφαρμογής του ελέγχου της ε, αλίας του γάδου. Το συζητήσαμε στις ε, κοινέ επιτροπές και δεν ξέρω αν γνωρίζετε τώρα η Γρυλανδία έχει ένα σχέδιο διαχείρισης και ο γάδος ε, παρακολουθείται πάρα πολύ καλά. Εκ πέραν αυτού υπάρχουν περιορισμοί, εποχικοί περιορισμοί, ποσοτικοί περιορισμοί και το Κοινοβούλιο ενημερώνεται απο, ε, για τα αποτελέσματα των κοινών ε, συνεδριάσεων των Επιτροπών κάθε χρόνο. Τώρα, όσον αφορά το κοκκινόψαρο, έγινε μία έκθεση αξιολόγησης. Ένα ζήτημα που προκύπτει είναι ότι η έκθεση αυτή η αξιολόγησης ολοκληρώθηκε το 2010, πριν την ανανέωση δηλαδή, και υπήρξε μια συμφωνία για, τον διαχειρισμό, για, την διαχείριση του, της αλίας του κοκκινόψαρου και η Ευρωπαϊκή Ένωση σκοπεύει να τηρήσει την συμφωνία της ε, NIAFC. Όσον αφορά τις νέες ρήτρε, όντως εισήχθησαν καινούργιες ε, ρήτρε. Εμείς το βλέπουμε ως κάτι πάρα πολύ θετικό. Και για μας εγγύεται την ε, επίτευξη βιωσιμότητας και βιώσιμης αλίας. Αυτά πολύ συνοπτικά για το κόκκινο ψαρό και θα σταματήσω εδώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Κανείς δεν ζητά το λόγο. Θα δώσω λοιπόν το λόγο στην κυρία Μάισνερ για τα συμπεράσματα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ όλους που συμμετείχαν σε αυτή τη συζήτηση. Σε γενικές γραμμές ε, παρατηρώ μια γενική συμφωνία. Φυσικά θα, υποστηρίξουμε τις προτάσεις της έκθεσης. Αρμοδι... Όσον αφορά την αρμοδιότητα, μας απάντησε ο συνάδελφος. Δεν έχω κάτι να προσθέσω και εγώ πραγματικά απορούσα γιατί η Επιτροπή Ανάπτυξης ήταν αρμόδια για αυτό, αλλά ε, Μάλλον αυτό οφείλεται στις υπερπόντιες χώρες και περιοχές. Το ζήτημα της υπεραλίευσης είναι πραγματικά πολύ σημαντικό. Πρέπει να προσέξουμε, παρότι δεν είμαστε η Επιτροπή Ελίας, αλλά πρέπει να προσέξουμε ως Επιτροπή Ανάπτυξης να προσέξουμε τι γίνεται σε αυτές τις χώρες. Δεν είμαι η Δήμων, ιδιαίτερα δεν είμαι η Δήμων στον τομέα της Αλίας όπως άλλοι συνάδελφοι, αλλά πραγματικά αναφέρθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι υπάρχει μια ενδεκτική ποσόστοση η οποία ελέγχεται και φυσικά πρέπει να ελέγχουμε εάν όντω υπάρχει αυτή η παρακολούθηση και αν είναι βιώσιμη η αλληλεία των ε, συγκεκριμένων ψαριών αυτών. Από πλευρά μας αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να υποστηρίξουμε την Επιτροπή Αλληλείας και να συμφωνήσουμε. Ευχαριστώ. Σας υπενθυμίζω ότι η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών λύγει την Τετάρτη, 19 Σεπτεμβρίου το μεσημέρι. Η ψηφοφορία στην Επιτροπή μας θα λάβει χώρα στις 9 Οκτωβρίου. Περνάμε στο σημείο 7 της ημερησίας διάταξης. Σημειωθείς από τα κράτη-μέλη πρόοδος προς την επίτευξη του στόχου της διάθεσης του 0,7% του ακαθάριστου εγχώριου εισοδήματο για την ανάπτυξη. Εφημισμό, βέβαια. Γιατί φοβούμε πω πρόοδο στην πραγματικότητα δεν έχει σημειωθεί. Ε, θα υποφεληθούμε της παρουσίας τριών εμπειρογνωμόνων, ε, μία από την Κομισιόν, ε, μία από την Concord και ενός εμπειρογνώμονα ε, ενό τρίτου εμπειρογνώμονα. Η Κομισιόν ε, μέσα Ιουλίου ε, δημοσίευσε την έκθεση της για το θέμα αυτό. Περιλαμβάνει την πρόοδο των κρατών μελών προς την επιτεύξη του στόχου. στόχο ο οποίο είχε αναλυθεί ήδη από τη δεκαετία του 70 από τον ΩΣΑ. Να φτάσουμε δηλαδή στο 0,7% του καθάριστου χώρου εισοδήματο για την αναπτύξη. Όμως τα στοιχεία του 2011 παρουσιάζουν μάλιστα υποχώρηση σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Επιπλέον έχουμε καινούριους στόχους προχρηματοδότηση, για παράδειγμα προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Τα αριθμητικά στοιχεία για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν μειωθεί το 2011 από 0,44% στο 0,42% του ΑΕ. Πρέπει εμείς να αξιολογήσουμε την επίδοση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ό,τι αφορά την ε, δημόσια ε, βοήθεια, ε, αναπτυξιακή βοήθεια. Η Κομισιόν έχει υποβάλει την έκθεσή της. Κυρία Ρενάτε, Χάλεν ε, θα μας την παρουσιάσει. Ο κ. Κάκενμπος θα μας αναφέρει τις βασικές γραμμές της έκθεσης Concord και η κυρία Ελιστον θα παρουσιάσει ε, τις, ε, τα στοιχεία που διαθέτει η ΟΑΝ. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσία τους τρεις εμπειρογνώμονες. Δίνω το λόγο στην κυρία Ρενάτε Άλεν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Χαίρομαι διότι θέσατε για άλλη μια φορά αυτό το σημαντικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Στην πρώτη διαφάνεια βλέπετε τον τίτλο, δηλαδή η έκθεση λογοδοσίας που υποβάλλουμε ετησίως αφορά την χρηματοδότηση της ανάπτυξης υπό την ευρεία έννοια. Και θα ήθελα να τονίσω ότι η χρηματοδότηση για την ανάπτυξη είναι κάτι πολύ περισσότερο από την παροχή κονδυλίων για την ανάπτυξη. Μας ενδιαφέρει λοιπόν... Μας ενδιαφέρουν όλα τα κεφάλαια που καλύπτονται από την ατζέντα των Ηνωμένων Εθνών μετά από το Monterey το 2000. Δηλαδή μιλάμε για όλους τους τομείς, την αρρωγή και την συνέργεια δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Επίσης μιλάμε για το διεθνές εμπόριο, για το διεθνές εμπόριο, τη ε, δημόσια ε, χρηματοδότηση σε διεθνές επίπεδο, το εξωτερικό χρέος και την αντιμετώπιση συστημικών ζητημάτων. Μιλάμε λοιπόν για το παγκόσμιο σύστημα συναλλαγών και η συνένεση του Μοντερέι το 2008 αντιμετωπίστηκε και από το γύρο της Ντόχα μέσα στα πλαίσια της χρηματοδότησης των κλιματικών αλλαγών, της ενέργειας του περιβάλλοντος και ούτω καθεξής. Πρόκειται για πολυσχεδή, ζητήματα και εστιάζουμε την προσοχή μας στην εποπτεία των όντα δηλαδή της επίσημης αναπτυξιακής αρρωγής. διότι εκτός από την Ευρωπαϊκή Ένωση κανένας άλλος φορέας δεν είχε ασχοληθεί με αυτό το θέμα. Μας ενδιαφέρει λοιπόν η απόδοση και αποτελεσματικότητα των κρατών μελών και της Κομισιόν σε αιτήσια βάση και υποβάλαμε αυτή την έκθεση τελευταία τον Ιούλιο. Η επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια δεν είναι η πιο σημαντική πηγή χρηματοδότησης, αλλά είναι βασική για τις φτωχότερες χώρες. Υπάρχουν μεμονωμένοι και συλλογικοί στόχοι αναπτυξιακής αρρωγής και θα ήθελα να σας τονίσω ότι η υπάρχει όλο ένα και διονγκούμενος ανταγωνισμός για να φτάσουμε στους αναπτυξιακούς στόχους. Αυτή τη στιγμή, και ως προς τα παγκόσμια, τα παγκόσμια δημόσια αγαθά. Τα επόμενα έτη θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το θέμα στα διάφορα διεθνή φόρα. Έχουμε τη διάσκεψη Ρίο συν 20 και μέσα στα πλαίσια των Ηνωμένων Εθνών θα γίνει συζήτηση για την βιώσιμη ανάπτυξη και μια στρατηγική χρηματοδότησης για τους βιώσιμους αναπτυξιακούς στόχους. Και η έκθεση θα υποβληθεί μέχρι το 2014 στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Και ως προς τις κλιματικές αλλαγές, τη στιγμή που η πρώτη φάση 10-12 φτάνει στο τέλος της, θα, θα προσπαθήσουμε να δώσουμε συνέχεια και αυτό αφορά και την ε, το 2020 καθώς και μεγαλύτερη χρηματοοικονομική κινητικότητα γενικότερα μέχρι το 2020. Από πλευράς ανάπτυξης θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι η βιώσιμη αναπτυξιακή ε, στόχη που είναι η ναυαρχίδα μας, η ναυαρχίδα των περιβαλλοντολόγων, μέσα στα πλαίσια της ατζέντα μετά το 2015, θα πρέπει να ενταχθούν σε αυτό το γενικότερο πλαίσιο. Και με βάση αυτά τα διεθνή δεδομένα θα πρέπει να αντιδράσουμε και προβήκαμε στη σύσταση μιας ομάδας και μιας υπηρεσίας για να ασχοληθεί με περιφαλλοντικά ζητήματα οικονομικά και με την ατζέντα μετά το 2015. Ελπίζουμε ότι όλα τα θεσμικά όργανα θα προσαρμοστούν με τη μεθοδολογία τους, διότι ε, υπάρχει ο φόβος ότι η επικέντρωση βρίσκεται αλλού και όχι σε μας ούτε στην ομάδα εργασίας του Συμβουλίου, ούτε σε επίπεδο επιτροπής. Δηλαδή, μας ξεπερνούν τα γεγονότα, με άλλα λόγια. Για να σας δείξω ότι η επίσημη αναπτυξιακή αρρωγή, η όντα, δεν είναι το πιο σημαντικό μέσο, ήθελα να σας δώσω αυτή τη γραφική παράσταση ε, μέσα στα πλαίσια της έκθεσης λογοδοσίας. Βλέπουμε ότι οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών είναι το μεγαλύτερο έσοδο των αναπτυσσόμενων χωρών και αυτό αφορά χώρες μέσου εισοδήματος. Η επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια θα πρέπει να διαδραματίσει πολύ σημαντικό ρόλο σε χώρες χαμηλού εισοδήματος, διότι εκεί πρέπει να έχουμε πρόσβαση και σε άλλους πόρους. Αυτή η γραφική παράσταση σας δείχνει ότι μας ενδιαφέρουν όχι μόνο οι εισρωές αλλά και οι εκροές από τις αναπτυσσόμενες χώρες μέσα στα πλαίσια των χωρών μεσαίου εισοδήματος. Ως προς την έκβαση του 2011 θα ήθελα να πω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν ο μεγαλύτερος δωρητής, η Ευρωπαϊκή Ένωση σε επίπεδο 27 το 2011 και εδώ βλέπετε σε σχετικούς και απόλυτους όρους τα συνολικά ποσά και ε, στην άλλη στήλη βλέπετε το μερίδιο του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος όπως ε, εξελίχθηκε μεταξύ 2002 και 2005 έχετε τις χώρες DAC ε, στην κόκκινη στήλη, ε, τα ε, μέλη των Ηνωμένων Εθνών είναι το πράσινο, η Ιαπωνία είναι το ΜΟΒ και ούτω καθαξής. Μιλάμε για χώρες δηλαδή DAC και εκτός DAC. αλλά μειώθηκε η επίσημη αναπτυξιακή αρρωγή της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε απόλυτους και σε σχετικούς όρους. Δεν θέλω να επαναλάβω πράγματα που γνωρίζετε, αλλά θα ήθελα να σας πω ότι η παγκόσμια βοήθεια έχει επίσης μειωθεί. Δεν αφορά δηλαδή μόνο την αποτελεσματικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά για μια παγκόσμια τάση όπως διαγράφεται μιλάμε για μείωση 400 εκατομμύριων ευρώ. Αλλά είμαστε πολύ μακριά από τη δέσμευση που είχαμε αναλάβει μέσα στα πλαίσια της στοχοθέτησης του 2015. Και θα βρισκόμαστε σε ένα επίπεδο 0,45 το 2015, δηλαδή θα χρειαστούμε 25 χρόνια επιπλέον για να φτάσουμε στο 0,7% που είχαμε ορίσει αρχικά. Επίσης υπάρχουν δεσμεύσεις στην Αφρική, δηλαδή θα πρέπει να προβούμε σε αύξηση 50% προς την Ήπειρο, αλλά εφόσον μιλάμε για ευθύνουσα πορεία δεν μπορώ να διαβλέψω ε, αυξήσεις ως προς την Ήπειρο της Αφρικής. Αν δούμε την περίοδο 2004-2011 είδαμε ότι είχαμε μια αύξηση 28% και ούτε το μισό δεν πήγε προς την Αφρική της επίσημης αναπτυξιακής αρρωγής. Υπάρχουν καλά και κανένα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 προσπάθησε να ανταποκριθεί στις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες. Δηλαδή, 0,15% χρηματοδότηση του ΑΕ, του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος δηλαδή εστιάζουμε την προσοχή μας στις πλέον ενδεείς χώρες μέσα στα πλαίσια της συνεργασίας. Και αυτή η τάση θα συνεχιστεί να υφίσταται και στο μέλλον μέσα στα πλαίσια της συγκεκριμένης στοχοθέτησης πολλά περισσότερα θα πρέπει να γίνουν για να φτάσουμε στη στοχοθέτηση του 2015. Δεν είμαι σίγουρη για το κατά πόσο μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο μέσα στα πλαίσια της χρηματοοικονομικής ε, ε λιτότητας την οποία υφιστάμεθα, αλλά η μείωση της χρηματοοικονομικής βοήθειας προς τρίτες χώρες δεν είναι η σωστή απάντηση. Όπως είπε και η Κομισιόν το Μάιο, το Συμβούλιο προετοίμασε την έκθεση του προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως προς την επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια για ε, μέσα στα πλαίσια δηλαδή της λογοδοσίας στο Συμβούλιο και η αρχηγοί μας προσπάθησαν να ανταποκριθούν, όχι ρητορικά, λέγοντας ότι θα προσπαθήσουμε να ανταποκριθούμε στη στοχοθέτηση μέχρι το 2015, άρα υπάρχει συνεχής δέσμευση των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων για να ανταποκριθούμε στις τάσεις που διαγράφονται μέχρι τούδε. Αυτή είναι και τελευταία διαφάνεια. Εδώ βλέπετε τι τις μεμονωμένες στοχοθετήσεις των κρατών μελών ως προς τους στόχους που θα πρέπει, τους οποίους πρέπει να φτάσουμε μέχρι το 2015. Θα δώσω τώρα το λόγο στους συναδέλφους από το Concord και το One. Um, θα σας ε, μιλήσω για την έκθεσή μας αλλά και θα απαντήσω και στην έκθεση που μόλις μας ε, παρουσίασε ο φίλος μου, ο συνάδελφός μου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, έχει δύο κομμάτια παρουσίασή μου. Στο πρώτο τμήμα θα αναφερθώ στο, στην έκθεση που μας ε, παρουσιάστηκε σε ιδιαίτερα ό,τι αφορά το ότι η επίσημη αντιξιακή αρρωγή δεν είναι η πιο σημαντική πηγή εισοδήματο και βοήθεια για αυτές τις Ε, θα μιλήσω για την εξασφάλιση χρηματοδότηση, για το χρέο κλπ. Ε, για σε ό,τι αφορά την ε, εσωτερική, την εγχώρια ε, κινητοποίηση των χρηματοδοτήσεων, αυτό είναι πολύ σημαντικό, πολύ σημαντικό χρηματοδότηση να γίνεται εγχώριο για να ξεφύγουν από την εξάρτηση και από τη φτώχεια. Ε, ο, οι για παράδειγμα, είναι το πιο καλό εργαλείο που διαθέτουν οι χώρες. Πλην όμως, ε, χρειαζόμαστε περισσότερες δεσμεύσεις ε, για ε, πιο δίκαια φορολογικά συστήματα, καθώς επίσης και να βοηθηθούν για να αποφύγουν την φοροδιαφυγή, την ε, αποχώρηση των κεφαλαίων κλπ. Παράνομες ροές και ε, φοροδιαφυγή ε, φτάνουν στο 1,5-3 εκατομμύριο δολάρια το χρόνο, ε, ευρώ το χρόνο. μας ανησυχεί όλο και περισσότερο το γεγονός ότι πολλές χώρες που στο παρελθόν είχαν εξασφαλίσει σταθερότητα στο χρέος ε, υποχωρούν εξαιτίας οικονομικής ε, κρίσης και εξαιτίας τη μείωσης της ενίσχυσής τους. Ε, χαιρόμαστε που αναλαμβάνονται δεσμεύσεις για να βοηθηθούν οι χώρες ως προς το χρέος τους και χαιρόμαστε που αναφέρεται η έκθεση και για τις για, την, για τον υπεύθυνο δανεισμό. Και έτσι οδηγούμε και στη, στις, ε, ε, στους καινοτόμους τρόπους δράσεως. Ε, θα πρέπει να δούμε ποιες είναι οι διαθέσιμες πλατφόρμες του blending, της ανάμιξης δηλαδή των ενισχύσεων, τα τελευταία χρόνια έχουμε δει ότι το ιδιωτικό χρέος είναι συνώνυμο του δημόσιου χρέους. Αυτό θα πρέπει να ε, φαίνεται λίγο λοιπόν σε οποιαδήποτε ανάλυση ανακούφιση του χρέους ε, και επίσης θα πρέπει και οι ενδιαφερόμενες χώρες να συμμετάσχουν σε αυτή τη διαδικασία του blending. Ε, δηλαδή της ανάπτυξης επίσημης και ιδιωτικής κρατικής και ιδιωτικής αναπτυξιακής αρρωγής. Τέλος, ε, χαιρόμαστε που η έκθεση υποστηρίζει τον ε, φόρο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, χρηματοοικονομικών συναλλαγών. Όμως ε, ε πιστεύουμε ότι ε, δεν θα δημιουργήσει σημαντικά ποσά αν δεν μείνουμε προσιλωμένοι στην χορήγηση επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας. Ο φόρος αυτός υποστηρίζεται από την κοινωνία των πολιτών αλλά θα πρέπει να συνδέεται με καινοτόμους τρόπους χρηματοδότησης ανάπτυξης και της κλιματικής αλλαγής της. Τώρα, για τη δική μας έκθεση, ε, τα ποσά είναι πολύ χαμηλά, η συνάδελφός μου θα μιλήσει γι' αυτό, αλλά πιστεύουμε ότι δεν συνδέονται τα λόγια με τις πράξεις, τα λόγια των κρατών μελών εννοώ με τις πράξεις, ε, του τι υπόσχονται με το τι πράττουν. Η δέσμευση είναι 0,7% αλλά χρειάζεται και δράση πλευρά των πολιτικών προκειμένου να επιτευχθεί το 2015. Αυτό το αναφέρουμε και στην έκθεση Aid Watch και στην έκθεση χρέους. Σε ό,τι αφορά την ποιότητα της ε, βοήθειας, ε, δεν έχουμε και εδώ πολύ πρόοδο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να λάβει τα ενία και χωρίς την Ευρωπαϊκή Ένωση το project αυτό θα περιθωριοποιηθεί. Φαίνεται σαν να είναι στάσιμο αυτή τη στιγμή. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να συμμετάσχει πιο δυναμικά. Επίσης, μας ανησυχεί και η εξασφα... ο στόχος ε, της ε, επίσημης αναπτυξιακής αρρωγής θα πρέπει να είναι ε, η... όχι ε, στόχοι που συνδέονται με την εξωτερική πολιτική, αλλά ο στόχο θα πρέπει να είναι η εκρίζωση τη φτώχεια. Η Eurotad ε, είδε, επίσης διαπίστωσε επίσης ότι πάνω από 60% των συμβάσεων ε, χωρίς επίσημης αναπτυξιακής εισαγωγής πηγαίνει στον ιδιωτικό τομέα και τα δύο τρίτα από αυτά σε πολυεθνικές εταιρείε. Συνεπώς θα μπορούσε ενδεχομένως να μειωθεί η επίσημη δεξιακή αρρωγή που δίδεται μέσω διεθνών ε, πολυεθνικών εταιριών υπέρ εθνικών εταιριών που με αυτόν τον ε, τρόπο θα κινητοποιήσουν και, και τον όλο μηχανισμό των χωρών. Ευχαριστώ. Καταρχάς ευχαριστώ πολύ την Επιτροπή Ανάπτυξης για την πρόσκληση. Είναι τιμή μας. Λοιπόν, η One είναι ένας οργανισμός υπεράσπισης. Έχει πάνω από 3 εκατομμύρια μέλη σε όλο τον κόσμο και εργαζόμαστε με κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο και προσπαθούμε να καταπολεμήσουμε τη φτώχεια, να επιφέρουμε αλλαγή και παρότι η επίσημη αναπτυξιακή αρρωγή δεν είναι η κύρια προτεραιότητά μας είναι εν τούτης κάτι πάρα πολύ σημαντικό για μας, ιδιαίτερα όσον αφορά την αρρωγή προς τις φτωχότερε χώρες. Από το 2006 κάθε χρόνο ε, κάνουμε μία άσκηση την ΑΜ. Φέτος επικεντρωνόμαστε στις υποσχέσει της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καταρχά, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρώπη είναι σίγουρα το, πιο, ε, το μεγαλύτερο οικονομικό μπλοκ που διαστηριοποιείται στο τομέα αυτό και δεύτερον μέσα στο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο αναπτύσσεται μια νέα ευκαιρία. Περίπου 27% της αναπτυξιακής χρηματοδότησης της ε, Ευρώπης πηγαίνει σε θεσμικά ιδρύματα και αν δεν, και αν δεν υπάρξει μια γενικότερη συμφωνία ανάμεσα στους διεθνείς οργανισμούς, τότε η κατάσταση για τις στοχότερες χώρες θα γίνει πιο δυσχερή. Όπως βλέπετε, στόχος μας είναι να σώσουμε την ε, βοήθεια αυτή, να εξοικονομήσουμε αυτή την βοήθεια. Έχουμε την ε, διάσκεψη στις 22 και 23 Νοεμβρίου για να οριστικοποιηθούν ε, οι λεπτομέρειες του πολιτούς δημοσιονομικού πλαισίου. ποια είναι η πρόκληση για εμάς. Γνωρίζουμε ότι, για παράδειγμα, υπάρχουν ανάμεσα σε 18 και 30 δισεκατομμύρια περικοπών που έχουν προταθεί από διάφορα κράτη-μέλη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε αυτές ε, τις ε, περικοπές. Γνωρίζουμε ότι η Ισπανία έχει προτείνει 30 δισεκατομμύρια σε περικοπές. Και κάποια άλλα κράτη-μέλη συζητούν περικοπές ακόμα μεγαλύτερες. Ο μέσος όρος που προκύπτει είναι, τα, είναι εκεί 18 έως 30 δισεκατομμύρια. Πιστεύω πως δεν έχουμε αντιμετωπίσει ποτέ μια παρόμοια κατάσταση με τόσο πολλές περικοπές. Γι' αυτό πραγματικά τους ε, επόμενους δύο μήνες κάνω έκκληση, επίγουσα έκκληση να προστατεύσουμε την, το ADA, αυτό, αυτή την αρρωγή. Και εσείς οι ευρωβουλευτές έχετε ακόμα πιο σημαντικό ρόλο εσείς πρέπει να υπογράψετε τη Συμφωνία για το πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο και αν ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέσει όρια, τότε θα βοηθήσει πάρα πολύ το, στόχος μα, το στόχο μας. Χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Σουηδία, η Γερμανία και οι κάτω χώρες είναι αυτές που επιθυμούν τις ε, μεγαλύτερες περικοπές και ξέρουμε ότι οι πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης ενδιαφέρονται «87.000 άνθρωποι, Ευρωπαίοι πολίτες μέχρι τώρα, έχουν υπογράψει την αίτηση. Τώρα, όσον αφορά την βοήθεια, η βοήθεια δεν δίδεται με τον ιδανικότερο τρόπο, παρόλα αυτά όμως είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Εδώ βλέπετε μία σύγκριση των δωρητών και των θεσμικών οργάνων. Σε τέσσερα επίπεδα. Όσον αφορά τα κριτήρια διαφάνειας και εκπαίδευσης, έχουμε πάρα πολύ καλή θέση. Σίγουρα υπάρχει, υπάρχουν ακόμα τομείς που χρήζουν βελτίωση. όμως πιστεύω ότι βρισκόμαστε σε πάρα πολύ καλό ε, δρόμο. Εδώ βλέπετε το κενό χρηματοδότησης της επίσημης αναπτυξιακής αρρωγής παγκοσμίω. Βλέπουμε τη διαφορά από την υπάρχουσα αρρωγή μέχρι το στόχο του 0,7% του ΑΕΠ. Ας δούμε ιδιαίτερα το κενό στη χρηματοδότηση για την Αφρική στη διαφάνεια που βλέπετε. Εδώ απέχουμε ακόμα περισσότερο από τον στόχο του 0,7%. Η μόνη ελπίδα που έχουμε ήταν η παρατήρηση μια μικρή αύξηση το 2011 τη αναπτυξιακή βοήθεια προ την Αφρική. Γιατί όμω είναι το, το δημοσιονομικό πλαίσιο τόσο σημαντικό. Αυτή εδώ, αυτό εδώ το γράφημα, στη διαφάνεια αυτή, μα λέει πώ η επίσημη αναπτυξιακή αρρωγή πηγαίνει μέσω των ευρωπαϊκών ε, θεσμικών οργάνων. Θα δείτε ότι ακόμα και για τα πολύ μεγάλα, για τα μεγάλα κράτη, για τη Γερμανία, για την ε, Γαλλία, τα ποσοστά δεν είναι μεγάλα. Τι ζητάμε. Πραγματικά στόχος μας είναι η προστασία του οργάνου αυτού και η παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας. Και βλέπουμε ότι και το EDF και το, και το DCI βρίσκονται σε κίνδυνο για το μέλλον. Και γιατί ασχολούμαστε με αυτό, γιατί προσπαθούμε να το σώσουμε, γιατί έχει αποτελέσματα. Έχουμε αυτά εδώ τα αποτελέσματα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα ήθελα να πω και στον συνάδελφο ότι πραγματικά θα επιθυμούσαμε πάρα πολύ να μιλήσουμε και σε πραγματικό χρόνο για τα αποτελέσματα της βοήθειας. θα, οι συζητήσει αυτέ θα είναι πάρα πολύ σημαντικές και θα μας βοηθήσουν να καταλάβουμε ακριβώς τι γίνεται και πώς μπορούμε να βελτιώσουμε αυτό που ήδη γίνεται. Το μήνυμα της παρουσίασης αυτής, με άλλα λόγια, είναι ότι θα θέλαμε να συνεργαστούμε τους επόμενους ε, δύο μήνες και εσείς οι ευρωβουλευτές είστε πάρα πολύ σημαντικοί, όχι μόνο ε, με την δυνατότητα και την ε, αρμοδιότητα που έχετε να υπογράφετε, αλλά και με τις διασυνδέσεις σας. Έχετε διασυνδέσεις με τις κυβερνήσεις σας. Είστε οι, οι κύριοι αντιπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις χώρες σας και πραγματικά μπορείτε να συνεισφέρετε και να φροντίσετε να δοθεί το μήνυμα όσο το δυνατόν εντονότερα. Και πραγματικά θα χαρούμε πολύ να συνεργαστούμε και με εσά και με όργανα όπω η Concord. Σας ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μας δώσατε να παρουσιάσουμε αυτή την έκθεση. Ευχαριστώ πολύ. Δίνω το λόγο στην κυρία Ντεκάιζερ. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω τους τρεις εμπειρογνώμονες για αυτό το σήμα κινδύνου το οποίο εξέπεμψαν και για τις μελέτες τους. Να κάνω μερικές παρατηρήσεις. Καταρχήν, συμμερίζομαι αυτή την αίσθηση επίγοντος. Στο Βέλγιο, στη χώρα μου, ε, ειδικά ε, μόλις πριν από δύο μέρες σε μια συζήτηση για τα δημοσιονομικά μας ανακοίνωσαν μείωση το 2012 ήδη ε, της αναπτυξιακής βοήθειας. Στην αρχή δεν το είχαμε πιστέψει, αλλά όταν στο πλαίσιο της ε, οικονομικής διακυβέρνησης ε, ε, είδαμε τις αυστηρές γραμμές που υπέδειξε η Κομισιόν, καταλάβαμε ότι χρειάστηκε να χρειαζόταν να παγώσουμε τον, ένα κομμάτι μάλλον του προπολογισμού ανθιακής βοήθειας. Στην αρχή ελέγχθη ότι πρόκειται για ένα πάγωμα, δεν πρόκειται για περικοπή, αλλά στην πραγματικότητα ε, η ανθιακή βοήθεια είναι θύμα της προσπάθειας να μην ε, ε, πειράξουμε τους μισθούς και τις συντάξεις. Στην πραγματικότητα όμως ε, το πάγωμα θα γίνει μείωση. Και το γεγονός είναι ότι η οικονομική διακυβέρνηση με αυτούς τους τρομακτικούς περιορισμούς που έχει μας οδηγεί αυτόματα στο να πούμε στους πολίτες μας ότι ε, η αναπτυξιακή βοήθεια μένει σε δεύτερο πλάνο. Θα πρέπει να κινητοποιηθούμε, σίγουρα, αλλά αν δεν, γίνει ε, γίνουν καλύτερα ε, γνωστά τα κοινωνικά προβλήματα όχι μόνο της ευρωπαϊκή Ένωσης αλλά και σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρόκειται να πετύχουμε τίποτα. Όσο παραμένουμε σε αυτό το πλαίσιο, είναι η φτωχή εναντίον των φτωχών. Η φτωχή των δικών μας χωρών εναντίον των φτωχών των τρίτων χωρών. Και αυτό το βλέπουμε καθημερινά. Σας ευχαριστούμε λοιπόν για αυτό το έγγραφο. Μια ερώτηση. Έχετε μια σειρά αποδείκτες στις εκθέσεις αποτελεσματικότητας, ποιότητας, ε, διαφάνειας κλπ. κλπ. Προφανώς δεν μπορούμε να, δεν έχουμε χρόνο να αναλύσουμε τον τρόπο με τον οποίο κάνατε τις μετρήσεις. Αλλά ήθελα να σας ρωτήσω, ε, αυτά τα στοιχεία τα έχετε δώσει στις κυβερνήσεις και ποια είναι η αντίδρασή τους. Το Βέλγιο, για παράδειγμα, ε, αναφέρεται επανειλημμένος με μάλλον αντικά στοιχεία παρόλο που ε, είμαστε πολύ δραστήριοι σε θέματα αναπτυξιακή ε, βοήθειας. Παρουσιάσατε αυτά τα στοιχεία στι κυβερνήσει. Euh, η Πρόεδρος, θέλω να κάνω και εγώ μερικά σχόλια. Με πολύ πάθος και σαφήνεια παρουσιάσετε τις εκθέσεις. Είναι σαφές ότι η μείωση από 0,44 στο 0,42 δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια αρχή. Τουλάχιστον αυτό είναι ο μεγάλος φόβος μας. Με την συνθήκη της Ένωσης που περιορίζει τα ελλείμματα στο 0,5% του ΑΕΠ ε, η πίεση στην αναπτυξιακή ε, βοήθεια θα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Και θέλω να χρησιμοποιήσω αυτή την ευκαιρία για να πω ότι όπως και πολλοί άλλοι εδώ και 15 χρόνια βλέπουμε αυτά που λέγαμε να γίνονται αλήθεια. Η... Γίνεται ε, όλο και πιο σημαντικό οι αναπτυσσόμενες χώρες να διατηρήσουν τους φυσικούς τους πόρους και θα ήθελα να ξεκινήσουμε μια εκστρατεία ε, που να καταδεικνύει πώς η πολυεθνικέ εταιρείε δεν πληρώνουν φόρους, ιδιαίτερου σε αφρικανικές χώρες όπου δραστηριοποιούνται και θα μπορούσαμε να εστιάσουμε σε ένα μηχανισμό τον οποίο χρησιμοποιούν εδώ και πολλά, εδώ και κάποια χρόνια, πολύ αποτελεσματικό, που ε, είναι τα υποπροϊόντα, συγγνώμη, τα παράγωγα προϊόντα, έτσι ώστε να μεταφέρουν τα κέρδη τους σε φορολογικούς παραδείσους. Με αυτόν τον τρόπο κρύβουν τα κέρδη τους και ε, φόρο αποφεύγουν ε, σε χώρες όπως η Τανζανία, το Μαλί, η Ζάμπια, η Νιγερία κλπ. Εδώ και περίπου 10 χρόνια προσπαθούμε να μας υποβάλλεται έκθεση αναχώρα Ε, δεν, δεν ήταν κάτι πολύ αυτό που ζητούσαμε, πλην όμως χάσαμε 10 χρόνια για να το καταφέρουμε. Θα πρέπει ταυτόχρονα να κινητοποιήσουμε και τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις, να διατηρήσουμε την πίεση σε ό,τι αφορά την επίσημη αναπτυξιακή αρρωγή, αλλά και ταυτόχρονα ο καθένας μας ε, να κάνει μία έρευνα για κάθε μία από τις πολυεθνικές και το τι μέσα χρησιμοποιεί για να αποφεύγει να φορολογείται στις χώρες του τρίτου κόσμου, στις αμψιόμενες χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται. Ο λόγος του κύριο Γκέρεντς. Ε, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Φοβούμαι ότι η Βερονίκ Κέζερ έχει δίκιο. Το Βέλιο δεν είναι μεμονωμένη περίπτωση. Εδώ βρισκόμαστε ενώπιον ενός σύριαλ, στο οποίο δίδεται συνεχώς συνέχεια. Και βλέπουμε ότι σε περίοδο ισχνών αγελάδων δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε αλλά αυτό αφορά και την περίοδο παχαίων αγελάδων. Δηλαδή δεν μπορούμε, μπορούμε να επιβάλλουμε στα κράτη-μέλη να τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους. Βλέπουμε ότι στο Σύμφωνο Σταθερότητας 60 υποδείξεις έγιναν, 60 φορές δεν βρέθηκε λύση. Φτάνουμε λοιπόν σε μια συλλογική ανευθυνότητα. Αυτός είναι ο φεντεραλισμός που προτείνεται. Όπως είπε και η Βερονίκ, υπάρχει επισφάλεια και στις χώρες δωρητές. Και πρέπει να αντιμετωπίσουμε και την εξωτερική πραγματικότητα. Βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη περίοδο. Καταρχήν δεν θα πρέπει να αποκλίνουμε από το στόχο του 0,7% δημόσια ε, επιδότη, δημόσιες ε, επιχορηγήσεις που αναλαμβάνουν τα κράτη. Θα πρέπει να είμαστε συνεπείς. Οι ροές αρρωγής θα πρέπει να ευεργετούν τις αναπτυσσόμενες χώρες και όχι το αντίθετο και τίποτα δεν θα πρέπει να μας μεταπίσει από αυτό το στόχο του 0,7%. Υπάρχει μεγάλη σιωπή από το Συμβούλιο. Ούτε ένα κράτος μέλος δεν έχει εκφραστεί επί του θέματος, ενώ πολλά μπορούν να υποθούν εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και θα ήθελα να κάνω μία έκκληση προς εμάς τα απειλητικά στοιχεία που διαγράφονται θέτουν σε κίνδυνο και τη συνενετική διαδικασία της Ένωσης. Εμείς θα πρέπει να διαφοροποιούμαστε. Δεν θα τηρήσουμε τους στόχους της χιλιετίας για την ανάπτυξη εάν δεν συνεχίσουμε με αυτή την πολιτική και δεν επικεντρώσουμε την προσοχή μας στις ε, χώρες που το χρειάζονται αμετάκλητα. Πώς θα εξηγήσετε στους Πορτογάλους που πρέπει να συνεχίσουν σε αυτή την προσπάθεια να χρηματοδοτήσουν τη Βραζιλία έτσι ώστε η Βραζιλία να δέχεται βοήθεια ενώ οι Πορτογάλοι στενάζουν και πρέπει να αναζητήσουν εργασία στη Βραζιλία. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε λίγο πιο συνεπείς, να μην αντιφάσκουμε. Και δεν πρέπει να έχουμε πατερναλιστική στάση έναντι των άλλων. Εγώ δεν είμαι καθόλου υπερήφανος από τις διαπιστώσεις που μας έδωσαν οι τρεις εισηγητές τους οποίους και ευχαριστώ. Εμείς τον Οκτώβριο, κατά τις ημερίδες ανάπτυξης, θα πρέπει να συγκεκριμενοποιήσουμε αυτούς τους στόχους. Δεν τολμώ καν να μιλήσω για τις ειδικέ χρηματοδοτήσεις για την μείωση των κινδύνων από τις κλιματικές αλλαγές. Το έχω πει μυριάδες φορές. Δεν έχει κανένα νόημα να μιλάμε θεωρητικά. Εκεί που έχουμε περιθώρια ελιγμού, ας είμαστε πιο συνεπείς για να κερδίσουμε σε, σε αξιοπιστία. Αξιοπιστία δική μας, η οποία άλλο ένα και υποσκάπτεται. Μαρτίνες. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι η έκθεση που μας υπέβαλαν οι φίλοι μας και ιδιαίτερα η έκθεση του Φορέα One που εγώ γνώριζα εδώ και καιρό. Τα στοιχεία αυτά είναι δραματικά, είναι διαφανή. Όλοι συνάδουν μαζί με τους συναδέλφους. Όλα συγκλίνουν. Εδώ είμαστε επτά παρόντες, έξι. Και όταν φύγω κι εγώ σε ένα λεπτό θα μείνετε πέντε. Δεν νομίζω ότι έχει νόημα να τα αναμοχλεύουμε αυτά μεταξύ μας. Η Ελοής είπε «Ελπίζουμε το κοινοβούλιο» κλπ. κλπ κοινοβούλιο, το κοινοβούλιο εκπροσωπεί τις κοινωνίες μας, τίποτα άλλο. Και στην τελευταία ακρόασή μας για την ανθρωπιστική βοήθεια και την ανάπτυξη το επαναλάβω. Το είπε και ο κύριος Γκέρενς και μίλησε για συνέπεια προπαντός. Δυστυχώς όμως έχει αλλάξει η διαδικασία ευρωπαϊκής οικοδόμησης. Επρόκειτο για ένα σχέδιο αλληλεγγύης μεταξύ μας, ενδοκινοτικά, όχι προς τα έξω. Και με βάση αυτή την αρχή της αλληλεγγύης θα έπρεπε να γίνει μια προβολή προς τα έξω. Δεν μπορούμε να, αγνοήσουμε ότι άλλαξαν τα πράγματα. Αυτή η αρχική αλληλεγγύη δυστυχώς εξέλιψε. Όταν ο κύριος Γκέρενς μιλά για συνοχή, συνέπεια, Σαρλ, το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει ενδοκινοτική συνοχή. Και δυστυχώς η μόνη συνοχή και συνέπεια είναι ότι κόβουμε τη βοήθεια προς τα έξω. Δηλαδή υπάρχει συνοχή των δυνάμεων και αλληλεγγύη των δυνάμεων του κακού και όχι του καλού. Σε μια κατάσταση κρίσης και επειδή μερικοί τη χρησιμοποιούν, τι κάνουν. Αποδομούν τα κράτη που ήταν αλληλέγγυα. Και αυτό συμβαίνει σε κάθε χώρα. Δεν μπορούμε να ζητάμε το αδύνατον ή κάτι από αυτόν που δεν μπορεί να το εκπληρώσει. Μιλάμε για συστήματα υγείας, εκπαίδευσης, συντάξεις, κοινωνικές υπηρεσίες. Μα οι κυβερνήσεις πώς θα ανταποκριθούν. Πώς μπορούμε να μιλάμε για 0,7% για διεθνή αλληλεγγύη. Μα υπάρχει εσωτερική ασυνέπεια. Γι' αυτό υπάρχει ασυνέπεια και προς τα έξω. Αυτή δυστυχώς είναι η πραγματικότητα που διέπει και το κοινοβούλιο μας. Γιατί δεν κινούμεθα κάπου στη στρατόσφαιρα. Εμείς εκπροσωπούμε πολιτικά αυτούς που εκπροσωπεί και το Συμβούλιο. Τέλος. Τι να περιμένουμε λοιπόν. Θα πρέπει να γίνει μια μεγάλη κινητοποίηση από εμάς και να αντισταθεί η κοινωνία. Αυτό που είπε και η Βερονίκ, γιατί οι πλέον φτωχοί στις χώρες μας αντιδρούν για λόγους αυτοσυντήρησης. Δηλαδή, ε, τι κάνουν, αντιτάσσονται στους φτωχούς που τους περιστοιχίζουν. Όπως είπε και ο Γκέρενς, τι θα κάνουμε με τους Πορτογάλους που συνεισφέρουν στην ανάπτυξη. Όχι μόνο επειδή οι νέοι θα πάνε στη Βραζιλία, οι νέοι από την Πορτογαλία, αλλά και από την Ισπανία και ίσως κάποια στιγμή και από το Λουξεμβούργο. Γιατί ζητούνται επενδύσεις, επενδύσεις δεν ζητάνε χρήματα από τη Βραζιλία, ζητάνε περισσότερα χρήματα για επενδύσεις στο εξωτερικό. Οι Βραζιλιάνοι δεν χρειάζονται χρήματα από την Κίνα για να υποστηρίξει την οικονομία τους. Θα πρέπει να εξορθολογήσουμε τη συζήτηση στο ακρόαση της προηγούμενης εβδομάδας ελέγχθησαν πολλά, αλλά μου σηκώθηκαν οι τρίχες όταν ένας από τους ομιλητές είπε ότι για κάθε ευρώ που δαπανούμε για να βελτιώσουμε τις σχέσεις μεταξύ ανθρωπιστικής πολιτικής και πολιτικής ανάπτυξης αποταμιεύονται επτά, μα μου σηκώθηκαν οι τρίχες πώς είναι δυνατόν να κόβουμε με το ψαλίδι και μετά να λέμε θα συνεργαστούμε. Και θα υπάρχει συνδρομή ανθρωπιστικής βοήθειας και αναπτυξιακής βοήθειας. Και για κάθε ευρώ που δίδεται θα μπορούσαμε να έχουμε αποταμιεύσει 7. Μα θα πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ τι λέμε σε σχέση με τους μηχανισμούς που χρησιμοποιούμε. Και όποιος βρίσκεται και επειδή βρισκόμαστε σε αυτή την κατάσταση, θα πρέπει η αρχή της αλληλεγγύης να είναι η κινητήριος δύναμή μας και θα πρέπει να διέπει όλες τις χώρες. Γι' αυτό θα πρέπει να καταβάλουμε υπεράνθρωπες προσπάθειες και σε Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Χωρίς να θεωρούμε ότι διαφέρουμε από το Συμβούλιο ή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι απότοκο όλων των άλλων. Είναι προέκταση όλων των άλλων. Εμείς δεν είμαστε μια διαφορετική οντότητα, δεν είμαστε οι καλοί της υπόθεσης. Εμείς οι έξι που είμαστε παρόντες, εμείς οι λίγοι. Αυτή είναι μια πραγματικότητα που πρέπει θεωρώ ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Εγώ στην ηλικία μου δεν μπορώ να μπω σε αυτή τη συλλογιστική, δηλαδή να παίρνουμε από εδώ κομματάκια, από εκεί κομματάκια. Δείτε τι γίνεται στην Ολομέλεια και ποιο προϋπολογισμό θα εγκρίνει η Ολομέλεια και πού θα γίνουν οι περικοπές. Γιατί ξέρουμε από πού θα γίνουν οι περικοπές. Πρόκειται για τους πιο αδύναμους κρίκους και αυτοί θα σπάσουν. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να κινητοποιηθούμε, να μιλήσουμε σε συμβιωτική σχέση με τις ΜΚΟ και ούτω καθεξής. Θα πρέπει να υπάρξει συνέργεια και συνέργειες, γνωρίζοντας όμως την πραγματικότητα την οποία ζούμε. Μη ζούμε εκτός πραγματικότητας είναι μισητή αυτή η πραγματικότητα. Αλλά για αυτήν φέρουμε ευθύνη και θα πρέπει να την μεταλλάξουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριος Βάγκελ. Έχει το λόγο. Έχουμε πολύ καθυστέρηση, λάβετε το υπόψη σας. Θα είμαι πολύ σύντομος. Συμφωνώ ότι η κρίση δημιούργησε ένα καινούριο πανόραμα. Είναι ελάχιστες οι χώρες ε, που οι κάτοικοι τους πιστεύουν ότι είναι πλούσιοι. Ακόμα και στις πιο πλούσιες χώρες ε, όλοι νιώθουν ότι γίνονται φτωχότεροι. Όλο και φτωχότεροι. Οπότε το κριτήριο της γενεοδορίας προς τους άλλους, της αλληλεγγύης και του ανοιχτού πνεύματος ε, για αυτούς που έχουν αναγκή αλλάζει. Αλλάζουν τα κριτήρια. Συνεπώς, η παρατήρησή μου είναι εξή. Μεταξύ άλλων επιχειρημάτων θα πρέπει να ε, δούμε και το πώς χρησιμοποιούνται τα χρήματα που δίνουμε. Γιατί εμείς αλλάζουμε, αλλά αλλάζουν και αυτοί που λαμβάνουν την ενίσχυση. Αλλάζουν δηλαδή, βελτιώνονται, φαντάζομαι, υποθέτω. Οπότε βλέπω να λείπει αυτό το επιχείρημα, ότι δηλαδή τα χρήματα τα οποία χορηγούμε επενδύονται σωστά και βελτιώνουν την κατάσταση στους τόπους που φτάνουν. Αυτά τα επιχειρήματα χρειάζονται. Ο... Δίνω ξανά το λόγο στους εμπειρογνώμονες και την εκπρόσωπο της ε, Κομισιόν για δύο λεπτά στον καθένα. Many thanks. Ευχαριστώ. Δεν θα σταθώ σε όλες τις παρεμβάσεις, μόνο μερικά σημεία για τον φόρο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών ελέγχθη ότι δεν οριοθετείται σαφώς. Η Επιτροπή υπέβαλε μία πρόταση. Η επίσημη θέση μας είναι ότι θα ενταχθεί στο επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Βεβαίως θα ήταν καλύτερα να υπάρχει σωστότερη οριοθέτηση, αλλά δεν μπορώ να το ε, προβάλλω αυτό εξ ονόματος Επιτρόπου Φίσερ. Ως προς την αποτελεσματικότητα της ε, αναπτυξιακής βοήθειας ε, χρειάζεται μεγαλύτερη, χρειάζονται μεγαλύτερες ηγετικές δυνάμεις, περισσότερες ηγετικές δυνάμεις και δεν θα ήθελα να μιλήσω για τις ε, παγκόσμιες δεσμεύσεις και υποχρεώσεις που έχουμε αναλάβει. Θα πρέπει να προβάλλουμε μία προστιθέμενη αξία, γιατί παρά τις υποχρεώσεις της προώθησης παγκόσμιας ατζέντα για την ε, βοήθεια και την ανάπτυξη, θέλουμε να ορίσουμε ένα πλαίσιο αναπτυσσόμενων χωρών, όπως είπε και ο κύριος Βάιγκελ, να δούμε δηλαδή πώς μπορούμε να υποπτεύσουμε καλύτερα αυτό το πλαίσιο, έτσι ώστε και οι χώρες να δαπανούν σωστά αυτά τα χρήματα. Επίσης, ως προς την λογοδοσία, υπάρχει και από πλευράς ε, δωρητού, όχι από, ε, από την πλευρά του ευεργετούμενου κράτους. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να μας απασχολεί στα πλαίσια της ευρωπαϊκής ατζέντα. Θα μπορούσαμε να κάνουμε ε, πολύ περισσότερα στη, στον κοινό προγραμματισμό της κατανομής της εργασίας. Και αυτό ιδιαίτερα για την ε, περίοδο μετά το 2013 και μετά το 2015, έτσι ώστε να κινηθούμε όλοι στην ίδια κατεύθυνση. Διακόπτη, Πρόεδρος. Θα είμαι σύντομο. Συμφωνώ. Οι περικοπές μόλις άρχισαν και θα ακολουθήσουν και άλλες. Το 0,7 λοιπόν δύσκολα θα το φτάσουμε χωρίς πολύ σοβαρή πολιτική διαβούλευση. Όμως είναι σημαντικό και ποτέ δεν ήταν πιο σημαντικό. Και πρέπει να προσέξουμε. Εάν μειώσουμε τις ε, παροχέ τουλάχιστον να αυξήσουμε την αποδοτικότητα όσον αφορά τις χώρες μεσαίου εισοδήματος που λαμβάνουν ε, αυτήν την αρρωγή, ίσως θα έπρεπε να κοιτάξουμε το μοντέλο εφαρμογής αυτών των χωρών, το πώς αποφεύγουν ε, ε, την φτώχεια, πώς συνεισφέρουν στην απαλυφή της φτώχειας και τι μπορούμε να αντιγράψουμε και να ακολουθήσουμε. Διότι η αναπτυξιακή πολιτική είναι ιδιαίτερα σημαντική στην απαλυφή της φτώχειας. Για παράδειγμα, βιομηχανική πολιτική, πολιτική φορολόγηση, ξεκάθαρου κανόνε για τον θεμητό ανταγωνισμό. Τώρα δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο για την αλληλεγγύη. Η αλληλεγγύη είναι κέριο σημείο της κοινωνίας που θέλουμε να δημιουργήσουμε. Τέλος. το Κοινοβούλιο πραγματικά πρέπει να βγάλει τον αγώνα αυτόν προς τα έξω. Συμφωνώ με αυτό και αυτό είναι κάτι που πρέπει να εκφράσουμε, που πρέπει να δείξουμε. Φυσικά το έγγραφο της Aid Watch συντάχθηκε με βοήθεια ε, των ε, διεθνών οργανισμών στις ε, διάφορες χώρες και φυσικά οι συζητήσεις λαμβάνουν χώρα και θα συνεχίσουν. Ευχαριστώ πολύ αυτά από μένα. Ευχαριστώ πολύ να απαντήσω σε ορισμένα από αυτά τα σημεία. Υπάρχουν ορισμένα επιχειρήματα στην έκθεση των δεδομένων γιατί, UA, γιατί η βοήθεια έχει προστιθέμενη αξία όταν ε, αποδίδεται συνετά. Αυτό που βρήκαμε εμείς είναι ότι όταν ε, εξηγεί τους πολίτες ακριβώς πόσο λίγο από τον εθνι... από ποσό, πόσο μικρό ποσό από τον εθνικό προπολογισμό ξοδεύεται για αναπτυξιακή βοήθεια, όταν τους το εξηγούμε, μας λένε πως πρέπει να δώσουμε περισσότερα. Και πραγματικά έχουμε και βίντεο, έχουμε και ντοκουμέντο αυτό σε βίντεο. Μιλήσαμε με ανθρώπους στο δρόμο και μας είπαν ακριβώς αυτό το πράγμα. Όπω είπε τώρα ο κύριο Γκόρεντ, σίγουρα στα πλαίσια του πολιτού δημοσιονομικού πλαίσιου είναι πολύ δύσκολο να γίνει. Πρέπει όμω να τονίσουμε στου αρχηγού ότι υπάρχει αυτή η ανάγκη. Ιδιαίτερα φέτο. η φετινή χρονιά είναι πάρα πολύ σημαντική και πρέπει να υπάρξει λογοδοσία, πρέπει να υποστηριχθούν οι παροχέ αυτέ. Όσον αφορά την ε, κυρία Ζολή και αυτό που είπε για του ίδιου ε, πόρου, συμφωνώ απόλυτα. Πρέπει να του προστατεύσουμε. Όμω η διαφυγή κεφαλαίου και η φοροδιαφυγή είναι πάρα πολύ σημαντικά ζητήματα. Αύριο το πρωί θα το συζητήσουμε στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων, μάλιστα, και θα παρουσιάσουμε και εκθέσεις και ελπίζω να ενδιαφερθούν οι ομάδες. Και πραγματικά κλείνοντας θα ήθελα να πω ότι ε, προσδοκώ τη συνεργασία σας. Είναι δύσκολο το ζήτημα, αλλά πραγματικά ελπίζω σε μια συνεργασία και στο ρόλο που μπορείτε να παίξετε εσείς οι ευρωβουλευτές. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και τους εμπειρογνώμονες μας για αυτή την εμπεριστατωμένη παρουσίαση. Τώρα θα στραφούμε στο σημείο 8 της ημερήσιας διάταξης, δηλαδή την σύναψη της Σύμβασης για την Φυσιστική Βοήθεια. Η συγητής είναι ο κύριος Ντέβα, ο οποίος όμως δεν είναι παρόν. Ο κύριος Μίτσελ τον αντικαθιστά. Η Επιτροπή μας ε, ενημερώνει σε τακτά χρονικά διαστήματα για την επαναδιαπραγμάτευση της επιστηστικής βοήθειας του 99 που είναι ένα μέσο, σημαντικό μέσο για να συνεισφέρουμε στην παγκόσμια διατροφική ασφάλεια. Επίσης, μέσα στα πλαίσια μιας επιπρόσθετης ε, πολιτικής ε, διατροφικής αρρωγής, θα πρέπει ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εγκρίνουμε το όλο πλαίσιο έτσι ώστε το Συμβούλιο να συμφωνήσει εξ ονόματος της Ένωσης πριν από το τέλος του Νοεμβρίου. Θα ήθελα ο κύριος Μίτσελ να μας μιλήσει για αυτό το σχέδιο συστάσεων. Well, σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Οχριό μπροστά στον κύριο Ντύρβα. Αλλά θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Μου ζήτησε να παρουσιάσω την έκθεση εκ μέρους του. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, ζητήθηκε να δώσει τη συγκατάθεσή του για αυτό για τη σύμβαση για την επιστηστική βοήθεια. Η σύμβαση του 1999 ήταν μια πολυμερή σύμβαση ανάμεσα στι ΗΠΑ, τον Καναδά, την Ιαπωνία, την Ελβετία, την Αυστραλία και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τέθηκε σε ισχύ την δεκαετία του 60 με σκοπό τον συντονισμό και την απαλυφή των γεωργικών πλεονασμάτων έτσι ώστε να βοηθηθούν οι χώρες που το, που το έχουν ανάγκη. Η συμφωνία αυτή έληξε τον Ιούνιο φέτος και συμφωνήθηκε να μην επεκτείνει την ε, σύμβαση αυτή, διότι είχαν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες για μια νέα σύμβαση. Η επαναδιαπραγμάτευση της σύμβασης ε, περιλάμβανε τον εξυγχρονισμό της, έτσι ώστε να υπάρχει καλύτερη ανταπόκριση στις επιστημιστικές ανάγκες του ε, φτωχού πληθυσμού. Αυτό πάει πέρα από την επιστημιστική βοήθεια, περιλαμβάνει και ανθρωπιστική βοήθεια και ε, περιλαμβάνεται στην ε, πολιτική ε, της, της ανθρωπιστικής βοήθειας. Τώρα, ο εισηγητής αναγνωρίζει ότι έχουν γίνει σημαντικές βελτιώσεις από την παλαιότερη σύμβαση για παράδειγμα, τώρα είναι ένα όργανο που προσανατολίζεται περισσότερο στους ε, αποδέκτες της βοήθειας. Επίσης, μεταφε... μεταλλάσσεται από μία προσέγγιση που εστιάζεται στα προϊόντα προς μία προσέγγιση που εστιάζεται στους ε, λήπτες. Περιλαμβάνει διάφορες επιχειρήσεις καθώς και παρεμβάσεις, επιστημιστικές παρεμβάσεις. Επίσης, δίδεται περισσότερη έμφαση σε λύσεις οι οποίες διευκολύνουν μια μετάβαση στην ε, εξυγίανση και ανάκτηση στα προγράμματα εξυγίανσης και ανάκτησης παρά της ε, απλής βοήθειας. Η νέα σύμβαση τονίζει την ανταλλαγή πληροφοριών και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών ανάμεσα στα συμβαλλόμενα μέρη, και αυτό θα επιτρέψει την ε, Επιτροπή να γίνει ένα περισσότερο ενεργό φόρουμ για, την, ε, για τον συντονισμό των δωρητών και την αμοιβαία μάθηση. Επίσης, στοχεύει στην ευ ευρύτητα και την διαφάνεια όσον αφορά τους ε, τα ενδιαφερόμενους, οι οποίοι ενδιαφερόμενοι θα προσκληθούν να συμμετάσχουν στην, ε, στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Επισητιστικής Βοήθειας. Επίσης, τα οι δυνατότητες βελτίωσης. Τα συμβαλώμενα μέρη μπορούν να κληθούν να δηλώσουν την ελάχιστη ε, βοήθεια που μπορούν να παρέχουν. Επίσης, θα, θα ασχοληθεί η νέα σύμβαση και με το τι γίνεται στην περίπτωση που καθυστερεί κάποια παράδοση της βοήθειας στις ε, χώρες που έχουν ανάγκη καθώς και της προσαρμογής ε, στις παγκόσμιες ε, τιμές των τροφίμων. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να συνεχίσει τις πιέσεις για μια εξυγχρονισμένη επιστημιστική βοήθεια, με την, κυρίως με την παροχή επιχορηγήσεων. Επίσης, πρέπει να βελτιωθεί ο συντονισμός με, μακροπρόθεσμες, ε, με μακροπρόθεσμο στόχο την βελτίωση της ε, γεωργικής παραγωγικότητας και των ε, εισοδημάτων των κατοίκων της υπαίθρου. Γι' αυτό έχουν, μπορούν να χρησιμοποιηθούν προγράμματα. Για παράδειγμα, το, το DCI, το Όργανο Αναπτυξιακής Συνεργασίας. Επίσης χρειαζόμαστε μία αμοιβαία δέσμευση ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών. Δυστυχώς όμως δεν υπήρχε η επιθυμητή συμμετοχή ορισμένων κρατών μελών. Η συνεχιζόμενη ανάγκη για επισητιστική βοήθεια είναι προφανής. Και ο εισηγητής πιστεύει ότι οι τροποποιήσεις που έγιναν σε σχέση με την προηγούμενη σύμβαση είναι ένα πολύ μεγάλο βήμα προς τα εμπρός. Γι' αυτό λοιπόν ο εισηγητής προτείνει το Κοινοβούλιο να δώσει τη συγκατάθεσή του. Τέλος, ο εισηγητής ελπίζει για μια ελάχιστη ετήσια δέσμευση για το 2013 και ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ενημερώνει να κρατά πλήρως ενημερωτό το Κοινοβούλιο για την πρόοδο της σύμβασης και σχετικά με το χρονοδιάγραμμα τώρα, η νέα σύμβαση μπορεί να τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου του 2013, εάν ε, την επικυρώσουν πέντε συμβαλόμενα μέρη μέχρι φέτος τον Δεκέμβρη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν η κινητήριος δύναμη πίσω από αυτήν την ανανέωση της σύμβασης. Και με το που δώσει τη κατάθεσή του το Κοινοβούλιο, τότε το Συμβούλιο θα μπορεί να προχωρήσει στην επίσημη ολοκλήρωση των ε, διαπραγματεύσεων της ανανέωσης ε, και το ιδανικό θα ήταν αυτό να γίνει μέχρι το Νοέμβριο φέτος, μέχρι τους επόμενους δύο μήνες. Και ελπίζω λοιπόν ιδανικά η Επιτροπή να υιοθετήσει στην Ολομέλεια του Οκτωβρίου και να ψηφίσει την νέα σύμβαση. Δεν, γίνεται, δεν είναι δυνατή κατάθεση τροπολογιών για την, για την για τα επιμέρους σημεία Τη νέα σύμβαση. Αυτά είχα να πω και χάρηκα πάρα πολύ που μπόρεσα να παρουσιάσω την έκθεση εκ μέρου του κυρίου Ντύρβα. Σας ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος. Τώρα θα δώσω το λόγο στην Κομισιόν, την κυρία Μαλόν, την εκπρόσωπο της Κομισιόν και τον κύριο Γκέρεντ πρώτα. Πρόεδρε, Έχω ένα σχόλιο και μία ερώτηση προς την Κομισιόν. Ο κύριος Ντέβα επιτέλεσε μία εξαιρετική εργασία. Και βλέπω ότι ένας πρώην υπουργός της Ιρλανδικής Δημοκρατίας μπορούσε να φτάσει, θα μπορούσε να φτάσει σε ένα τέτοιο αποτέλεσμα όπως έφτασε ο κύριος Ντέβα. Ε, αυτό που βλέπουμε ο, αυτό που, όπως βλέπουμε, πέντε θα πρέπει να προσυπογράψουν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρείται ένας προσυπογράφων ή θα μπορούσαν να συμμετάσχουν μονομένα τα κράτη-μέλη. Αυτό από τεχνικής πλευράς είναι ερώτηση. Θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι για το Νοέμβριο, όπως είπε και ο κύριος Μίτσελ. Η κυρία Μαλόν. Τρία λεπτά τρία λεπτά κατά το μέγιστο. Για να απαντήσω στον κύριο Γκέρενς, η Food Assistance Convention, η σύμβαση αυτή επισχιστικής βοήθειας, αποτελεί μια πραγματικά μεικτή συμφωνία, δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να συμμετάσχει στη σύμβαση και κάθε κράτος μέλος ε, κατά συνέπεια, καθώς και η υποψήφια χώρα η Κροατία μπορούν ε, μεμονωμένα να προσυπογράψουν. Εάν λοιπόν Έχουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση συν τέσσερα κράτη-μέλη που έχουν κυρώσει τη συνθήκη στις 30 Νοεμβρίου. Μέχρι τις 30 Νοεμβρίου θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Πρώτου 2013. Θα θέλαμε όλα τα μέρη, διαπραγματευτές ΗΠΑ, Καναδάς, Ιαπωνία, Αυστραλία, Ευρωπαϊκή Ένωση και Ελβετία να είναι έτοιμη για εν ώψη της προθεσμίας της 30ης ε, Νοεμβρίου. Θα πρέπει να κυρωθεί λοιπόν μέχρι τότε η σύμβαση. Παράλληλα ενθαρρύνουμε τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συμμετάσχουν στη νέα σύμβαση. Γιατί όπως είπε και ο εισηγητής, η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν η κινητήριος δύναμη της Σύμβασης του 1999 και για μας είναι πολύ σημαντικό να συνεχίσουμε και να δείξουμε ότι δεσμευόμαστε για να μην υπάρχει πια ε, επισητιστική ανασφάλεια προς τους, ε, ως προς πλέον φτωχούς και θα πρέπει να το επιδιώξουμε άμεσα. Η νέα σύμβαση αποτελεί βασικό στοιχείο απόδειξης της αλληλεγγύης μας των πιο ευάλωτων από τον, χωρών από τον τρίτο κόσμο. Κύριε Μίτσελ, θέλετε να μας μιλήσετε για τα συμπεράσματα. Ε, είναι Πολύ συχνά οι Βρετανοί αναθέτουν αρμοδιότητε σε ανώτατου Ιρλανδού αξιωματού κυβερνητικού. Με πολύ χαρά το κάνουμε αυτό. Εκχωρούμε αρμοδιότητε. Ε, ε, ευχαριστώ πολύ τον κύριο για την, την παρατήρησή του. Ελπίζω, ε, την παρατήρησή του. Ελπίζω πράγματι να προχωρήσει αυτό. Ευχαριστώ. Ωραία. Χαίρομαι που το σημειώνετε. Κύριο Γκέρνς, θέλει ξανά το λόγο. Νομίζω ότι αυτό έχει σχέση με τι αρμοδιότητε του Κοινοβουλίου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Για το θέμα τη ε, επικύρωση. Αν το Κοινοβούλιο δεν επικυρώσει. Τι σημαίνει αυτό, αν η συμφωνία αυτή επικυρωθεί από ένα κράτος μέλος, μετράει για την θέση σε ισχύ. Γιατί το Κοινοβούλιο έχει δικαίωμα να μπλοκάρει αυτή τη συμφωνία. Σύμφωνα με τη χάρη στη συνθήκη Λισαβόνας. Οπότε αυτή η ιστορία ότι πρέπει να είναι πέντε κράτη-μέλη δεν μου αρκεί. Θα ήθελα να είμαστε σαφείς σε αυτό. Υπάρχουν δύο διαφορετικά θέματα. Πρώτον, το κείμενο της καινούρια σύμβασης που αναφέρει ότι θα τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2013 αν πέντε μέρη την έχουν επικυρώσει μέχρι τη 30 Νοεμβρίου. Αυτό το αναφέρει η σύμβαση. Τώρα το άλλο θέμα είναι ένα εσωτερικό νομικό ζήτημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάτι τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων τα μέρη, κάτι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισαν ότι θέλουν ένα πραγματικό μεικτό διεθνές, ε, ε, ένα πραγματικό μεικτό διεθνή μηχανισμό. Δηλαδή Ευρωπαϊκή Ένωση και κράτη-μέλη μαζί να επικυρώσουν την καινούρια σύμβαση. Αυτή ήταν μια καινούργια ε, ιδέα. Ε, έχουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα 15 κράτη-μέλη, συν την Κροατία, που έχουν όλοι τη δυνατότητα να υπογράψουν την καινούργια σύμβαση. Δεν είναι μία υπογραφή. Αν το κοινοβούλιο αποφασίσει να μην δώσει τη σύμφωνη γνώμη του, αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα επικυρώσει την καινούρια σύμβαση. Οπότε, ποια είναι η κατάσταση. Η κινητήρια δύναμη πίσω από τη σύμβαση που έχει ένα πολύ σημαντικό έγγραφο πολιτικής που αναφέρεται σε αυτή τη σύμβαση και που είναι ένας από τους μεγαλύτερους χρηματοδότες, δότες ε, τέτοιου είδου βοήθεια, δεν θα μπορέσει να υπογράψει αυτή τη σύμβαση την οποία τόσο δραστήρια διαπραγματεύτηκε. Ευχαριστώ. Ε, Πολύ ωραία. Θα πρέπει να περάσουμε στο σημείο 9. Όμως η τη Κομισιόν δεν είναι παρούσα, οπότε προτείνω να περάσουμε στο 10. Γνωμοδότηση Μίτσελ για τον προπολογισμό σημείο 10 της ημερησίας διάταξης. Στις 3 Σεπτεμβρίου η, προ, ε, ψηφίσαμε τις ε, τροπολογίες μας για τον προπολογισμό του 2013. Η τελευταία, το τελευταίο στάδιο θα είναι να ψηφίσουμε τη γνωμοδότηση που ε, συνοδεύει αυτές τις τροπολογίες και εκφράζει την θέση της Επιτροπής μας για τις ε, δημοσιονομικές προτεραιότητες του επόμενου χρόνου. Κύριε Μίτσελ, ακριβώς αυτό το σχέδιο γνώμης θέλω να μας ε, παρουσιάσετε. Ε, κύριος Μίτσελ, μια και η γνώμη θα ψηφιστεί αύριο, θα επαναλάβω γιατί το έχω, έχω ήδη ξαναπεί, ορισμένες από τις ε, σημαντικότερες ανησυχίες μας σε ό,τι αφορά τη διαπραγμάτευση με το Συμβούλιο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ευθύνη εναντί των αναπτυσσόμενων εταίρων της. Τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και τα κράτη-μέλη έχουν αναλάβει δεσμεύσει να καταπολεμήσουν την φτώχεια στον αναπτυσσόμενο κόσμο και θα πρέπει να τη στηρίσουμε. Τα στοιχεία έφτασαν καθυστερημένα αλλά το έχουμε πει τόσο πολύ και τόσες πολλές φορές. Ε, ένα από τα βασικά σημεία του κειμένου είναι η αντίθεσή μας στις προτάσεις του Συμβουλίου να κόψει παραπάνω από 50 εκατομμύρια ευρώ σε αναλήψη υποχρεώσεων και 150 εκατομμύρια ευρώ για τις ε, ε, πληρωμές του, του μηχανισμού χρηματοδότησης. Αυτό δημιουργεί προβλήματα στην υγεία, την εκπαίδευση, στην ασφάλεια των τροφίμων που είναι τομείς κλειδί για να πετύχουμε τους στόχους της χιλιετίας. Επίσης, η χρηματοδότηση για την αντιμετώπιση του προβλήματος της κλιματικής αλλαγής θα πρέπει να είναι καινούργια και πρόσθετη. Επίσης, οι μειώσει στη χρηματοδότηση των τοπικών αρχών και των τοπικών φορέων επίσης δημιουργεί προβλήματα. Ε, αναφέρουμε το Ιράκ, το Ιράν, την Παλαιστίνη, το Αφγανιστάν και την Ιεμένη ιδιαίτερως ε, διότι τέτοιου είδους ε, περικοπές, ειδικά για αυτές τις χώρες, δεν είναι αποδεκτές αυτή τη στιγμή, διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει παίξει πολύ σοβαρό ρόλο στην σταθεροποίηση αυτών των περιοχών τα τελευταία χρόνια. Τέλος, εκφράζω την χαρά μου για το έγγραφο εργασία τη Επιτροπή Προπολογισμού σε ό,τι αφορά τη θέση του Συμβουλίου για το σχέδιο προπολογισμού του 2013, που δείχνει αυτό το έγγραφο ότι ο εισηγητής λαμβάνει υπόψη τι ανησυχίε μα, τέρους τις ε, ανησυχίες μας που αφορούν τις μειώσεις, τις περικοπές προτείνει το Συμβούλιο στην Αναπτυξιακή Βοήθεια. Δεν θα σας καθυστερήσω άλλο, δεν θα μας καθυστερήσω άλλο. Ε, το έχουμε επανειλημμένο συζητήσει το θέμα και ξέρω ότι η Επιτροπή συμμερίζεται τις απόψεις μου. Ευχαριστώ. Ε, το λόγο έχει Επιτροπή ο κύριος Κάρλο Άιλ, ο οποίος απουσιάζει. Υπάρχει κάποιος άλλος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που θα ήθελε να λάβει το λόγο. Ευχαριστώ. Επειδή δεν είναι ο υπεύθυνο, εδώ θα ήθελα να πω ότι συμφωνώ με την παρουσίαση, δηλαδή η Επιτροπή συμμερίζεται τις ανησυχίες του εισηγητή και θα ήθελα να πω ότι ήδη στο παρελθόν λέγαμε ότι ο προϋπολογισμός λαμβάνει υπόψη τους δικαιούχους πρωτίστως. Και νομίζω ότι ανταποκριθήκαμε σε αυτό το στόχο. Κύριε Μίτσελ, θέλετε κάτι να προσθέσετε. Όχι. Χαίρομαι που μας υποστηρίζει η Επιτροπή γιατί υπάρχουν συγκεκριμένες ε, στοχοθετήσεις και όταν φτάσουμε στην ώρα της ψηφοφορίας θα εκφράσουμε την απόψή μας. Ωραία, σας ευχαριστώ. Περνάμε τώρα στο προηγούμενο σημείο αν έχει φτάσει αν έχει φτάσει ο υπεύθυνο από την Επίτροπη. Όχι, περιμένουμε τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το σημείο υπαριθμών 9. Ωραία. Σημείο 9 της ημερήσιας ε, διάταξης, οι τοπικές αρχές στην ανάπτυξη. Ο κύριος Μπάλιο έχει το λόγο. Μάλλον φτάνει τώρα. Η Επιτροπή έχει συντάξει μία γνωμοδότηση προς περιφερειακές και τοπικές αρχές. Η Επιτροπή αποφάσισε την έναρξη μίας διαβούλευσης με τους εμπλεκόμενους φορείς. Και η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι το Δεκέμβριο 2012 με την συνεργασία των ε, τοπικών αρχών στην Ευρώπη αλλά και στην Αφρική και στη Λατινική Αμερική καθώς και στην Ασία σε συνεργασία με την πλατφόρμα το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Τοπικών Αρχών για την Ανάπτυξη. Επίσης θα συμμετάσχουν εμπειρογνώμονες για τη συνεργασία και την ανάπτυξη. Ο κύριος Μπάλιο που είναι επικεφαλής ε, της ε, Γενικής Διεύθυνσης ΔΕΦΚΟ έχει το λόγο για να μας παρουσιάσει τα βασικά σημεία του εγγράφου. Ευχαριστώ. Ζήτω συγγνώμη που καθυστέρησα. Αλλά αντιδρώ με βάση παυλοφικά καθαρά ενάψματα και βρέθηκα στο απέναντι κτίριο. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να σας ε, παρουσιάσω τις προτεραιότητες μας ε, ως προς τις, ε, τη συμμετοχή των τοπικών αρχών για το 2013. Όπως γνωρίζετε, το 2010-2011 άρχισε διάλογος με τις τοπικές αρχές και εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών και φτάσαμε στη δήλωση της Βουδαπέστης όπου οι οργανώσεις αυτές συμφώνησαν για να λάβουμε υπόψη περισσότερο τις τοπικές αρχές και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Ο Επίτροπος Πίμπαλξ ασχολήθηκε με τις τοπικές αρχές και τους εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών και στη συνέχεια υποβάλαμε δύο ανακοινώσεις. Πρώτον ως προς το ρόλο της κοινωνίας των πολιτών που εγκρίθηκε από την Επιτροπή την προηγούμενη εβδομάδα και στη συνέχεια είχαμε μια δεύτερη ανακοίνωση για το ρόλο των τοπικών αρχών. Πρόκειται για δύο διαφορετικούς φορείς, διότι η κοινωνία των ε, πολιτών απορρέει από ε, ιδιωτικούς φορείς, ενώ οι τοπικές αρχές αφορούν μια γενικότερη θεσμική πλαισίωση. Δηλαδή πρόκειται για διακυβερνητικό, κυβερνητικό καθαρά πλαίσιο. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν εστιάζουμε την προσοχή μας στους διάφορους φορείς που διαδρούν πώς θα αρχίσει η διαβούλευση αυτή για την προετοιμασία της ανακοίνωσης. Όπως είπε και η Πρόεδρος, προβλέπουμε μία σειρά διαβουλεύσεων κατά το τελευταίο τρίμηνο του έτους με εκπροσώπους των τοπικών αρχών που θα οδηγήσουν σε συστάσεις οι οποίες θα ληφθούν υπόψη για την προετοιμασία της ανακοίνωσης. Θα θέλαμε να συζητήσουμε κατά τις διαβουλεύσεις οκτώ σημεία τα οποία προετοιμάστηκαν στο έγγραφο αυτό που λάβατε. Το πρώτο αφορά το ρόλο των τοπικών αρχών στις ε, διεθνείς, στα διεθνή φόρα και εδώ μιλάμε για τον ρόλο των τοπικών αρχών. Θα θέλαμε όμως να το δούμε με τους εμπλεκόμενους φορείς, να δούμε δηλαδή πώς μπορούν οι τοπικές αρχές να συνδράμουν. Στη συνέχεια θέλουμε να ασχοληθούμε με την χρηστή διακυβέρνηση και το τοπικό εδαφικό επίπεδο. Όπως ξέρετε, οι τοπικές αρχές διαδραματίζουν σημαντικό θεσμικό ρόλο που ορίζει ο νόμος στις περισσότερες περιπτώσεις και αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να τονίσουμε τη χρηστή διακυβέρνηση σε επίπεδο διοικητικών περιφερειών. Θέλουμε να εμβαθύνουμε αυτό το θέμα. Έπειτα υπάρχει το θέμα της ε, εδαφικής ανάπτυξης, το οποίο συζητήθηκε μεταξύ εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών μέσα στα πλαίσια ενός καλώς διαρθρωμένου διαλόγου. Θέλουμε να δούμε τον εδαφικό χαρακτήρα που απομακρύνεται από την εγκάρσια προσέγγιση και να αντιμετωπίσουμε το θέμα τομεακά έτσι ώστε να έχουμε μια ολιστική προσέγγιση και καθαρά εγκάρσια, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις εδαφικές ε, ενότητες. Και θα θέλαμε να προωθήσουμε το διάλογο. Η αποκέντρωση είναι το τέταρτο σημείο. Ξέρετε ότι προωθούμε εδώ και χρόνια μία πολιτική αποκέντρωσης. Έχουμε διαθέσει 800 εκατομμύρια, αλλά το θέμα αυτό δεν είχε συζητηθεί με τις τοπικές αρχές αλλά μόνο σε επίπεδο κυβερνήσεων. Και εδώ θα θέλαμε να συνομιλήσουμε με τις τοπικές οργανώσεις ζητώντας μια ανάληψη υποχρεώσεων στα πλαίσια αποκεντρωμένων κρατών. Το πέμπτο σημείο που θα θέλαμε να συζητήσουμε αφορά την ε, προβληματική, τη συλλογιστική του αστικού χαρακτήρα των πόλεων. Μιλάμε για, μεγάλες, ε, για μεγάλα αστικά κέντρα, κάτι το οποίο επηρεάζει την ποιότητα ζωής των πληθυσμών. Και κατά συνέπεια οδηγεί στην απερίμωση πολλών περιφερειών, καθαρά αγροτικών περιφερειών. Θα θέλαμε λοιπόν να ε, γνωρίζουμε τις εμπειρίες αυτών των ε, φορέων για να δούμε πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις μεγαλοπόλεις ιδιαίτερα έναντι των αγροτικών περιοχών. Ο ρόλος των ε, τοπικών αρχών υπάρχουν φορείς στα πλαίσια των τοπικών αρχών και πολλές χώρες δυστυχώς δεν έχει ενισχυθεί ο ρόλος τους. Θέλουμε να δούμε πώς λοιπόν μπορούμε να υποστηρίξουμε και να ενισχύσουμε αυτές τις οργανώσεις. Τέλος, το έβδομο σημείο αφορά τις ε, δυνατότητες και το δυναμικό των τοπικών αρχών διότι οι τοπικές αρχές έχουν, διαθέτουν θεσμικό ρόλο παροχής υπηρεσιών προς τον πληθυσμό, αλλά δυστυχώς στις χώρες εταίρους υπάρχουν μεγάλες αδυναμίες ως προς την δράση των φορέων. Θα θέλαμε να το δούμε με τους άμεσα ενδιαφερόμενους για να γνωρίζουμε τι υποστήριξη μπορεί να δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αν τη ζητηθεί. Το τελευταίο θέμα αφορά μία συζήτηση με τους εμπλεκόμενους, βασικούς εμπλεκόμενους φορείς για να δούμε τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την ενίσχυση των τοπικών αρχών είτε σε επίπεδο κρατών καθαρά. για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στην παροχή υπηρεσιών προς τους πληθυσμούς. Αυτά τα θέματα θέλουμε να συζητήσουμε κατά το τρέχον τρίμηνο, έτσι ώστε να μπορέσουμε να υποβάλουμε μία πρόταση πολιτικής υφής που θα υποβάλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και είμαι στη διάθεσή σας για να απαντήσω σε τυχόν ερωτήσεις και να ρωτήσω κατά πόσο κράτη θέλουν να συνδράμουν σε αυτή την προσπάθεια. Ευχαριστώ για αυτή την παρουσίαση της ε, δράσης που προβλέπει η Κομισιόν για το ρόλο των τοπικών αρχών στην ανάπτυξη. Σημειώνω ότι δεν έχει ξεκινήσει, ε, βρίσκεται στο στάδιο της επεξεργασίας της. Το λαμβάνουμε υπόψη. Ε, Θα περάσουμε στο σημείο 21 της ημερήσιας διάταξης. Σας είχα αναφέρει εξ αρχής μια αλλαγή στην, στη σειρά Τα κοιτούσα και δεν μου δείξατε ότι θέλετε να πάρετε το λόγο. Όταν ζητάμε το λόγο συνήθως σηκώνουμε το χέρι μας. Εντάξει, εντάξει. Ασφαλώς και έχετε το λόγο. Δυστυχώς όμως χωρίς μικρόφωνο. Δεν μας ρωτήσατε αν θέλουμε να μιλήσουμε, γι' αυτό το λόγο δεν σήκωσα και εγώ το χέρι μου, Πρόεδρε. Λοιπόν, χαίρομαι που η Επιτροπή μας ε, προγραμμάτισε μια συζήτηση για τη θέση των τοπικών αρχών στην πολιτική ανάπτυξη ως βουλευτές. Πρέπει να συμμετάσχουμε σε αυτή τη συζήτηση που ως τώρα ήταν αποκλειστικό έργο της Κομισιόν. βλέπω ότι ακόμα και σήμερα δεν υπάρχει πολύ ενδιαφέρον από άλλου ευρωβουλευτές. Μόνο εγώ είμαι εδώ. Μετά το 2008 περάσαμε στην, σε πιο ψηλή ταχύτητα. Πολύ πρόσφατα διοργανώθηκε ο διαρθρωμένος διάλογος. Για ένα χρόνο διοργανώθηκαν σεμινάρια σε όλα τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα σε συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών και τις ε, τοπικές αρχές για να συζητήσουμε αυτό ακριβώς το θέμα. Ήταν λοιπόν επίγον και η Επιτροπή μας να ασχοληθεί. Γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά ότι είναι πρωταρχικής ε, σημασίας η συμμετοχή να είναι όσο πιο πλατιά γίνεται για να πετύχουμε τους αναπτυσιακούς στόχους της διεθνούς κοινότητας. Χωρίς την υποστήριξη των τοπικών αρχών που στην πλειοψηφία τους παρέχουν βασικές υπηρεσίε όπως η υγεία και η εκπαίδευση, τα αποτελέσματα των πολιτικών μας για την κατά τη ε, θα είναι φτωχά. Το... Οι άξονες της δράσης Κομισιόν υπογραμμίζουν το πώς είναι παράγοντες κλειδί οι τοπικές αρχές στους δύο βασικούς τομείς προτεραιότητας της ε, αναπτυξιακή μας πολιτικής. Η, ε, η διακυβέρνηση και η ανάπτυξη χωρίς εξαιρέσεις, χωρίς αποκλεισμούς. Ε, οι τοπικές ε, αρχές ε, έτσι κι αλλιώς εγγράφονται σε ένα πλαίσιο πολυτομιακό και οριζόντιο. Οι τοπικές αρχές συμμετέχουν στον σχεδιασμό των πολιτικών σε εθνικό επίπεδο και μερικές φορές και στις διαπραγματεύσεις συνεργασίας με τα διεθνή όργανα. Βρίσκονται λοιπόν κοντά στον πολίτη, έχουν δημοκρατική νομιμοποίηση και οι τοπικές αρχές ε, ενθαρρύνουν τις, ε, τη δημιουργία εταιρικών σχέσεων είτε δημόσιο ιδιωτικού τομέα είτε δημόσιο τομέα με τους πολίτες του. Με λίγα λόγια, η πρόσφατη ε, δήλωση για την αποτελεσματικότητα της ενίσχυσης συνοψίζει πολύ σωστά το ρόλο των τοπικών αρχών ως ενδιάμεσο ανάμεσα στους πολίτες και το κράτος, ε, έτσι ώστε να έχουν δημοκρατική βάση τα αναπτυξιακά προγράμματα. Αν η Κομισιόν αποδείξει το σημαντικό ρόλο των, εθνικών, των τοπικών αρχών στην υλοποίηση των στόχων της πολιτικής ανάπτυξης, τότε θα μπορέσουμε να ενισχύσουμε αυτή την προστιθέμενη αξία. Το έγγραφο όμως ε, δεν κάνει προτάσεις για καινούριες με συνεργασίας και βοήθειας ε, που θα μπορούσαμε να χορηγήσουμε στις τοπικές αρχές. Ε, θα ήθελα να πω βέβαια ότι ε, θα μπορούσαν ε, οι συγγραφείς του εγγράφου αυτού, μια και δεν εξέφραζαν την άποψη της ε, Κομισιόν, επίσημα της να πάνε πολύ πιο μακριά. Και θα ήθελα και εμείς να τους ενθαρρύνουμε. Θα ήθελα να ζητήσω από τους συναδέλφους να, να λάβουν την ευθύνη τους, όταν ψηφιστεί, κάθε φορά ψηφίζονται ε, μηχανισμοί αναψυχιακής βοήθειας, στην ψηφοφορία αυτή, αν ψηφίσουμε την τροπολογία 370, θα δώσουμε τη δυνατότητα στον συνάδελφο Μπέρμαν να διαπραγματευτεί με το Συμβούλιο για να αυξηθεί η χρηματοδότηση των τοπικών αρχών και θα επιτραπεί στην Κομισιόν να υλοποιήσει τις καλές προθέσεις που εκφράζει το έγγραφο μας παρουσίαση. Ευχαριστώ. Merci beaucoup. Je redonne la parole, Ξαναδίνω το λόγο στην Επιτροπή για να απαντήσω τον κύριο Τυρολιά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον κύριο Τυρολιά για την υποστήριξή του. Θα ήθελα να πω ότι τα κύρια θέματα που αναφέρθηκαν θα αποτελέσουν αντικείμενο συζητήσεων του επόμενου τριμήνου και με βάση στα συμπεράσματα θα υποβάλουμε προτάσεις στην ανακοίνωση μέσα σε ένα συνενετικό πλαίσιο. Ευχαριστώ. κυρία Γκρέσ, αύριο θα Τελικά αύριο θα έρθει. Άρα, σε αντίθεση με αυτά που σας προανακοίνωσα, δεν θα εξετάσουμε σήμερα την έκθεση ε, Γκρέσε για την βιοπειρατεία. Θα προσπαθήσουμε αύριο μετά την ψηφοφορία στην, ε, στις τροπολογίες του DCI να δούμε αν μπορέσουμε ε, να εντάξουμε αυτή την έκθεση. Διαφορετικά, αν υπερβούμε το χρόνο μας, ε, θα, θα το εντάξουμε κάπου αλλού, γιατί είναι κρίμα να το παρουσιάσουμε και ενώπιον δύο βουλευτών. Άρα τελείωσαν οι εργασίες, οι σημερινές μας εργασίες. Αύριο θα συνεδριάσουμε στις 10 εδώ και οι συντονιστές θα ε, συνέλθουν εδώ στις 9 το η ώρα για τους συντονιστές, 10 για την Επιτροπή σας. Ευχαριστώ, γεια σας.